Mes chers collègues, bonjour. Αγαπητοί συνάδελφοι, εσείς εκεί πίσω στην αίθουσα, καθίστε παρακαλώ. Ελάτε, καθίστε. Monsieur Robert Zille, on va commencer. Θα αρχίσουμε. Avant de commencer nos travaux. Προηγουμένως, πριν ξεκινήσουμε τι εργασίες μας για τη δέσμη μέτρων, θα ήθελα να χαιρετήσω στην αίθουσα την παρουσία εκπροσώπων της ομοσπονδία τη Ευρωπαϊκής Μεταφορών, όπου εκπροσωπούνται συνδικαλιστέ ε, οδηγοί φορτηγών από την Πολωνία, την Ρουμανία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο κλπ. Καλώς ήρθατε λοιπόν όλοι σας στην Επιτροπή μας. Θα συζητήσουμε λοιπόν σήμερα το μεσημέρι τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα. Και αρχίζουμε με τον χρόνο ανάπαυσης. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Φαντεκάμπ, και στη συνέχεια στον κύριο Μπαχ που δεν έχει φτάσει ακόμα. γιατί είναι εισηγητής της Επιτροπής Απασχόλησης και μετά στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές που θέλουν να εκφραστούν αφού έχουμε ακούσει τους διάφορους σκιώδεις εισηγητές. Τέλος θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο κύριος Λιζό πάντα πιστός στο πόστο του να μας δώσει την άποψη της Επιτροπής και μετά ο εισηγητής για τα συμπεράσματα. Κύριε Βίμ Φαντερ Κάμπ, λοιπόν, σας ακούμε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι σε πολύ καλή διάθεση Το δικό μου θέμα που έχει να κάνει με τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης έχουμε προχωρήσει πολύ. Δεν ε, έχουμε εξαντλήσει το θέμα και αύριο το πρωί θα έχουμε μια συνάντηση των ε, σκιωδών εισηγητών τη παρουσία ε, του εισηγητή γιατί είναι σκιώδες εισηγητές αλλά επιτρέπεται να είναι και ο εισηγητής αυτός καθεαυτός. Και στη συνέχεια θα εξετάσουμε το φάκελο μαζί με τον εισηγητή για το καμποτάζ, τον κύριο Ερτούγκ και για την απόσπαση εργαζομένων της κυρίας Κιλόνεν. Οι τρεις μαζί λοιπόν έχουμε αναλάβει τα θέματα τα εμπορικά και τα κοινωνικά. Τώρα έχω διάφορα σημεία στον κατάλογό μου και θα αρχίσω με τα ελαφρά εμπορικά οχήματα για τα οποία συζητήσαμε με τους σκιώδεις εισηγητές. Και είπαμε ότι είναι αυτά που είναι πάνω από 2,4 τόνοι και που κάνουν διεθνείς μεταφορές. Θέλουμε λοιπόν να τα συμπεριλάβουμε και αυτά, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει η επικουρικότητα. Οπότε, κάθε όχημα το οποίο προβαίνει σε διεθνείς μεταφορές και είναι 2,4 τόνοι ή περισσότερο, ε, συμπεριλαμβάνεται και μπίπτει στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού αυτού. υπάρχουν εξαιρέσεις για τον οικοδομικό τομέα. που έχει προβλήματα με το θέμα των μεταφορών. Το επόμενο θέμα μου έχει να κάνει επίσης με εξαιρέσεις. Πρόκειται για επιχειρήσεις και λεωφορεία που δεν έχουν τις μεταφορές σαν κύρια απασχόληστε. Πρόκειται για τραυλικούς, για φουρνάριδες ή τέτοια επαγγέλματα που χρησιμοποιούν τις μεταφορές αλλά δεν είναι η κύρια απασχόλησή τους. Οπότε και εκεί υπάρχει εξαίρεση όσον αφορά τον χρόνο ανάπαυσης, απασχόλησης κτλ. Επόμενη παρατήρηση. Στην αιτιολογική σκέψη θα πρέπει να αναφέρουμε κάτι και για τα οχήματα που οδηγούνται αυτόματα, δηλαδή χωρίς οδηγό. Ε, βλέπετε ο χρόνος τρέχει και οι εξελίξεις οι τεχνολογικές επίσης. Οπότε πρέπει να δούμε ο οδηγός τι είναι για τις περιπτώσεις τέτοιων οχημάτων Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό για να δούμε πώς θα το εξετάσουμε. Τώρα, πόσο χρόνο μπορεί να είναι στο δρόμο ο οδηγός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τρεις εβδομάδες και μετά πρέπει να επιστρέφει σπίτι του. Εγώ πρότεινα, επειδή έχω στην ομάδα μου πολλούς συναδέλφους από την Ανατολική Ευρώπη, τέσσερις εβδομάδες εκτός έδρας αλλά θα δούμε αύριο το πρωί που θα καταλήξουμε στην συνάντηση που θα έχουμε. Πάντως κάπου εκεί θα είναι τρεις ή τέσσερις εβδομάδες η περίοδος αναφοράς. Και αυτό συνδέεται βέβαια και με την ανάπαυση στην, ε, στο φορτηγό μέσα. Είναι και αυτό το οποίο συζητιέται πάρα πολύ στην Ανατολική Ευρώπη και υπάρχουν πολλές και διάφορες εμπειρίες. Οπότε θα ήθελα εδώ να καταλήξουμε σε κάτι συγκεκριμένο. Η ανάπαυση μέσα στο φορτηγό απαγορεύεται βάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πρόσφατη απόφασή του. Όμως εφόσον ο οδηγός θέλει ανάπαυση μέσα στο φορτηγό του αλλά σε ένα χώρο πάρκινγκ ανάλογο, εξοπλισμένο κτλ τότε μπορεί δύο, τρει το πολύ τέσσερι περίοδου σύντομη ανάπαυση 24 ώρων να μπορεί όντω να τις έχει μέσα στο φορτηγό του. Αυτό θα μπορούσε να λύσει ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Το βλέπω και στην Ολλανδία που όλο και περισσότεροι οδηγοί που καταλήγουν ένα Σαββατοκύριακο σε ένα, στο πάρκινγκ ενός βενζινάδικου τρώνε, ε, κατουράνε και δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς εκεί στα δέντρα, στο βουνό δίπλα στο Βεζινάδικο. Ενώ αν πρέπει να πάει στο ξενοδοχείο το Σαββατοκύριακο αυτός ο οδηγός φορτηγού, αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Πώς θα γίνει αυτό, φανταστείτε να έχουμε 55 τέτοια φορτηγά μεγάλος πανικός. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Δηλαδή ναι μεν να μην κοιμούνται μέσα στα φορτηγά τους, εκτός από την περίπτωση που μπορούν να παρκάρουν σε έναν χώρο κατάλληλα εξοπλισμένο. Ε, υπάρχει το θέμα των 45 ωρών ανάπαυση, αλλά και εδώ έχουμε βρει έναν συμβιβασμό το κατά πόσο... Συγγνώμη, ε, μιλάμε για την μικρή ανάπαυση των λεπτών, 45 λεπτών, που μπορεί να είναι 3 φορές 15 λεπτά. Και μετά ερχόμαστε και στις περιπτώσεις του φέρι και του τρένου. Γιατί αν είναι πάνω σε ένα φέρι, πάνω σε ένα τρένο το φορτηγό, τότε μπορεί κανεί, ο οδηγό δηλαδή, να κοιμάται. Μπορεί να μην είναι ιδεώδει οι συνθήκε, αλλά μπορεί να έχει ανάπαυση πάνω στο φέρι, πάνω στο τρένο με το φορτηγό του. Τώρα για τις τρεις ή τέσσερις περιόδους, τις τρεις ή τέσσερις εβδομάδες, αν δηλαδή ο οδηγό πρέπει να επιστρέφει σπίτι του κάθε τρεις εβδομάδες ή κάθε τέσσερις εβδομάδες. Και τι εννοούμε σπίτι το εννοούμε εκεί όπου κατοικεί. Η συζήτηση γίνεται και το κατά πόσο πρέπει να επιστρέψει εκεί που είναι η έδρα τη επιχείρησή του. Ναι, αλλά αν είσαι οδηγό, εγώ, και δουλεύει για μια δανέζικη εταιρεία, ε, δεν σημαίνει ότι κάθε τρει εβδομάδε πρέπει να επιστρέφει στην Κοπεχάγη, θε να πα στην οικογένειά σου. Οπότε θα πρέπει ε, να μπορεί να το κάνει αυτό και μπορεί να υπάρχει και η εξαίρεση άμα θέλει να πάει και διακοπές στην ε, παραλία της Ταραγώνας ας πούμε. Αυτό που δεν είναι λογικό είναι να του απαιτούμε να πάει στην έδρα της επιχείρησής του, στη Δανία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, η, η μεταφορά, ε, λεωφορεία δεν μπορεί να συγκριθεί με τα containers και τα συνδικάτα θέλουν ειδική ρύθμιση για τον ε, κλάδο των λεωφορείων. Έπειτα ερχόμαστε και στο θέμα του εφιού σταχογράφου. Όλο ο φάκελο του καμποτάζ, της απόσπασης και του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης μπορεί να ισχύσει μόνο εφόσον η εφαρμογή γίνεται καλά και σωστά. Γι' αυτό και πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να εγκαθιδρύσει όσο γίνεται πιο γρήγορα τους ευφυείς ταχογράφους. Η δικιά μου εμπειρία είναι ότι αν προτείνει ξεκάθαρη νομοθεσία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε η αγορά θα ακολουθήσει. Αν λέμε μ, οι ευφυείς ταχογράφοι 24, 26, 28 θα ισχύσουν, τότε τίποτα δεν θα έχουμε. Δεν είμαστε σαφείς δηλαδή για το πότε πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν. Πρέπει να πούμε 1η Ιανουαρίου 2020 για παράδειγμα. Αυτό πρέπει να είναι το χαρτί που θα παίξουμε στο Συμβούλιο. Σίγουρα είναι μια μεγάλη δυσκολία για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να καταλήξει σε ημερομηνία. Ελπίζω να μας ακούσει γιατί εν πάση περιπτώσει κάπως πρέπει να προχωρήσει και αυτό να πάρει. Δεν μπορεί χρόνο-χρόνο να καθυστερούμε. Δεν έχω την αίσθηση ότι 8 Ιουνίου θα έχουμε κάτι συγκεκριμένο από το Συμβούλιο, η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Μακρόν και όλοι οι υπόλοιποι θέλουν, λένε, να προστατεύσουν τον κλάδο των μεταφορών. Ναι, αλλά πρέπει να αποφασίσουν και τι θέλουν. Εντάξει. Μια που έχω το λόγο, μπορώ να τα πω κι αυτά, ότι θα έρθουν και εκλογές. Και μέχρι τις εκλογές φοβάμαι ότι ο καθένας ε, θα κάτσει πάνω στις δάφνες του και δεν θα προχωρήσει. Δεν είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Για τους ευφύς ταχογράφους, λοιπόν, πρέπει να προβλέψουμε και τεχνικά δηλαδή, να μπορεί ο ταχογράφος να καταγράφει από μόνος του και πότε διασχίζει τα σύνορα ένα φορτηγό. Πρέπει επίσης να υπάρξει, το είπαμε με τον ε, κύριο Ερτού και την κυρία Κιλόνεν, ότι θα ετοιμάσουμε ένα κεφάλαιο και το έχουμε ετοιμάσει ουσιαστικά για την ε, επεξεργασία των ε, τριών αυτών φακέλων. Και θέλω ήδη από τώρα να ευχαριστήσω τη γραμματεία, να, τους δύο που κάθονται εκεί στην άκρη από τη γραμματεία, γιατί τελικά κατάφεραν και έβαλαν στο χαρτί αυτό το κεφάλαιο. Και τώρα θα εκνευριστεί φυσικά το Συμβούλιο όταν θα δει πώς εμείς αντιμετωπίζουμε και πώς προστατεύουμε τα κοινωνικά δικαιώματα των οδηγών φορτηγών. Γιατί δεν πρόκειται εδώ πέρα μόνο για την ευελιξία, όπως το θέλει το έλξη στις μεταφορές, πρόκειται και για κοινωνική προστασία όπως την θέλει και η ομάδα των σοσιαλιστών και της ΓΚΟΕ είναι ένα ξεκάθαρο κεφάλαιο στο οποίο έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία έχοντας συνεργαστεί με τις εθνικές αρχές που έχουν αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, δεν θα φτιάξουμε καινούριο κέντρο στοιχείων, δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν, ούτε και σε σχέση με την προστασία των δεδομένων, αλλά πάση περιπτώσει έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία από τα κέντρα που συγκεντρώνουν δεδομένα. Οπότε, σας εξήγησα πώς έχουν τα πράγματα. Έχει ήδη δημοσιευθεί αυτό το κεφάλαιο. Όχι ακόμα, όχι. Ε. Δεν έχει Ωραία. Περιμένουμε να ξέρουμε και πότε θα ψηφίσουμε. Φαντάζομαι ότι θα μας ανακοινωθεί αυτό. Αυτά. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμ Βαντεκάμπ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, οπότε ζητώ συγγνώμη αγαπητοί ισχυώδεις συζήτητες, δεν θα έχετε 15-20 λεπτά όπως ο Θα είμαι λίγο πιο αυστηρός μαζί σας. Ωραία. Κυρία Ντεμόντε, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Βαντεκάμπα για τη σκληρή δουλειά που έκανε για τις συμβιβαστικέ και για την ευαισθησία του σε κοινωνικά θέματα που μας είναι και μας προσφυλή. Ευχαριστώ τους σκιώδεις, όλους όσους συνεργάστηκαν ε, στενά αυτούς τους μήνες. Πρέπει να πω ότι έχουμε καταλήξει σε κάποια σημεία σύγκλησης ε, μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις. Παραμένουν φυσικά και κάποια σημεία που χρειάζονται ακόμα δουλειά. Αύριο έχουμε μια νέα συνάντηση σκιωδών ε, όπου πιστεύω θα μπορέσουμε να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα. Όσον αφορά την ουσία των διαφόρων συμβιβαστικών είμαι υπέρ της εξαίρεσης ε, για τον ταχογράφο ε, για οχήματα μέχρι 3,5 τόνους για τις μεταφορές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός κράτου μέλους αρκεί να υπάρχει δυνατότητα το κράτος αυτό να εφαρμόζει τον πιο αυστηρό κανόνα ε, των 2,4 τόνων. Αντίθετος, ε, είμαι υπέρ του να διατηρηθούν οι 2,4 τόνοι για την εξαίρεση σε περίπτωση μεταφορά μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών μελών. Επίσης είμαι υπέρ, όπως είπε ο εισηγητή, για την εξαίρεση για τον τομέα των ε, οικοδομών. Πιστεύω ότι όσον αφορά τη μεταφορά με την κύρια δραστηριότητα του οδηγού, ε, εκεί η διατύπωση χρειάζεται να την ξαναδούμε. Όσον αφορά την ανάπαυση εντός του θαλάμου είναι ένα καθοριστικό θέμα και πολύ ευαίσθητο. Εκεί υπάρχει δικογνωμία μεταξύ των ομάδων και μεταξύ των αντιπροσωπιών. Πρώτα απ' όλα, ε, το διάστημα εβδομαδιαίας ανάπαυσης ε, θα πρέπει να σχετίζεται με τις αντισταθμιστικές περιόδους με μειωμένη εβδομαδιαία ανάπαυση που πρέπει να είναι στο σπίτι πιστεύω. Όταν λέμε σπίτι εννοούμε τον πραγματικό τόπο μονίμης κατοικίας. Ώστε να ξαναβρίσκουν και τις οικογένειές τους. Δεν ε, γίνεται δηλαδή να γίνεται εντός του φορτηγού. Επίσης θα πρέπει να βρούμε ένα συμβιβασμό όσον αφορά την επιστροφή στο σπίτι και πότε πρέπει να γίνεται. Μετά θα πρέπει να δούμε και τις απαιτήσει των πιο περιφερειακών περιοχών όταν το φορτηγό μεταφέρεται πάνω σε ένα τρένο ή σε ένα ε, Φεριμπότ. Ε, γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία. Η ψηφιακό ταχογράφο όσον αφορά τον έξυπνο, το δεύτερη γενιά δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε retrofitting το ταχύτερο δυνατόν. Τοποθέτηση δηλαδή. Με πιο αυστηρέ προδιαγραφέ. Με ε, καταγραφή σε πραγματικό χρόνο τη θέση του Ισδαλίκα. Διαφωνώ να υπάρχει δυνατότητα ότι δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το φορτηγό. Είναι δυνατό με, τη... με τις συσκευές που έχουμε ήδη στα χέρια μας. Αυτός ο τοχογράφος θα πρέπει να καταγράφει αυτόματα τη διέλευση από τα σύνορα. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν θα πρέπει να καταγράφεται στο πρώτο σημείο που αυτό είναι δυνατόν. Κάτι τελευταίο όσον αφορά τη μεταφορά ανθρώπων, επιβατών και εγώ συμφωνώ, πρέπει αυτούς τους δύο τομείς να τους διατηρήσουμε τους. Υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσει που αιτιολογούν διαφορετική εφαρμογή της ευελιξίας. Θα πρέπει μάλιστα να έχουμε εντελώ ε, διακριτές διατάξεις. Ευχαριστώ και πάλι για την επικοδομητική του συνεργασία του συναδέλφου και τον εισηγητή και ελπίζω ότι αύριο θα καταφέρουμε να βρούμε συμφωνία και στα σημεία που απομένουν. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντεμόντε. Κύριε ε, Ζήλε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Καρίμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Βήμ για τη δουλειά που έχει, κάνει, καθώς ε, και τους ε, άλλους εισηγητές, διότι μιλάμε για δέσμη μέτρων. Αυτά βέβαια δεν σημαίνουν ότι θα συμφωνήσουμε με όλα. Από πλευράς του ECR, όσον αφορά τις ελάχιστες απαιτήσει όσον αφορά την ε, ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε σχεδόν 500 ε, ε, τροπολογίες και έχουμε καταλήξει σε 70 θέματα συζήτησης. Πάντως εγώ θα αναφερθώ σε πέντε από αυτές. Όσον αφορά το LCV είμαστε κατά, διότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι ε, πρέπει να προσέξουμε ότι κάποια φορτηγά την καθίστανται από ελαφρά οχήματα για να μην χρειάζεται να τηρούν τους χρόνους ανάπαυσης. Ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όμως ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι συχνά ακόμα και διασυνοριακές μεταφορές πραγματοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, επιστροφή στον τόπο κατοικίας. Και πάλι θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βίμ που προσπαθεί να καταλήξει σε μια λύση όσον αφορά τον ορισμό αυτόν ε, για τον οποίο κανένας δεν γνωρίζει τι ακριβώς ε, σημαίνει. Ε, ζούμε στην ελεύθερη Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να μετακινούνται όπως θέλουν. Και να μην συγκρίνω την Ευρωπαϊκή Ένωση με την Σοβιετική Ένωση αλλά είχαμε ένα τραγούδι τότε που έλεγε ότι η διεύθυνσή μου δεν είναι το σπίτι μου, η πόλη μου, είναι η Σοβιετική Ένωση. Κάθε οδηγό λοιπόν μπορεί να επικαλεστεί κάτι τέτοιο, ε, να έχουμε έναν ε, βούλγαρο οδηγό. Ε, λέτε ωραία, πρέπει ο βούλγαρο να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ε, έτσι λοιπόν υποχρεούται ο οδηγό να επιστρέψει από τι Βρυξέλλε στην Βουλγαρία, αλλά μπορεί η οικογένειά του να μένει στην Ισπανία ή αλλού. Έτσι λοιπόν ε, επιβάλλεται ε, σημαντικό κόστος στον εργοδότη στην Κοπεχάγη για παράδειγμα για να στείλει πίσω τον οδηγό και μπορεί ο εργοδότης στην Κοπεχάγη, να πει ε, να σε απολύσουμε και να μείνει στο χωριό σου στη Βουλγαρία. Ποιος θα νοιαστεί για αυτόν τον φτωχό κύριο ή την κυρία. Κάποιο στις Βρυξέλλες ή κάποιο στην Κοπεχάγη θα, ασχοληθεί με την τύχη αυτού του ανθρώπου. Ας ε, γνωρίζουν οι πολιτικοί λοιπόν τι θέλουν να κάνουν εδώ. Χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία ο οδηγός ε, θα πρέπει να ενημερώνει τον εργοδότη που θέλει να περάσει τον ελεύθερο του χρόνο μετά από τις τέσσερις αυτές εβδομάδες. Δεν ε, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφερόμαστε σε συγκεκριμένο τόπο, διότι τι είναι ο τόπος διαμονής στο κάτω-κάτω. Επίσης, ε, ο χρόνος ανάπαυσης στην καμπίνα του οδηγού. Ε, ο χρόνος ανάπαυσης δεν επιτρέπεται να ε, πενιέται μέσα στην καμπίνα και έχουμε απόφαση του δικαστηρίου που δεν επιτρέπει μείωση του χρόνου ανάπαυσης. Με την συμβαστική πρόταση αυτή λοιπόν ε, ακολουθείτε την επιχειρηματολογία της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με μια τροποποίηση. θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ίδια ε, επιστοποίηση των ε, χώρων στάθμευσης σε κάποια κράτη-μέλη. Δεν θέλω να δημιουργήσουν τέτοιου ε, χώρους στάθμευση, διότι έτσι δημιουργείται ανταγωνισμός. Θα είμαι σύντομος. Δύο τελευταία τις παρατηρήσεις, έχουμε τον χρόνο οδήγησης. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε 180 ώρες ανά τέσσερις εβδομάδες, λαμβάνοντας υπόψη και τη θέση των πιο περιφερειακών χωρών. Και συχνά βλέπουμε εξελίξει. μπορεί σύντομα να δούμε νέα είδη ταχογράφων και έτσι κάποιε επιχειρήσει να χρειαστεί δύο φορέ να αλλάξουν ταχογράφου, το οποίο δεν θα θέλαμε να συμβεί. Σα ευχαριστώ κύριε Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Τζασίν Μέσνερ που είναι η συγκήτρια για την έκθεση αυτή δεν μπόρεσε να έρθει. Και εγώ θα μιλήσω εκ μέρους της. Όσον αφορά τα ελαφρά οχήματα και τη συμπερίληψή τους στον κανονισμό, αν υπάρχει πρόβλημα με τις διεθνείς μεταφορές αυτών των οχημάτων, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό θα πρέπει όσα είναι κάτω από 3,5 τόνους να έχουν εφή ταχογράφο εφόσον είναι σε διεθνείς μεταφορές. Αυτό προτείνουμε λοιπόν στον εισηγητή πώς θα ελεγχθεί το όχημα το οποίο ε, περνάει τα σύνορα ή δεν τα περνάει. Όσον αφορά την ανάπαυση μέσα στο φορτηγό, ακούσαμε τι είπε ο εισηγητής για να επιτρέπεται η ανάπαυση μέσα στο φορτηγό εφόσον αυτό παρκάρει σε χώρους που είναι εξοπλισμένοι κατάλληλα. Θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος όμως μέχρι να εγκριθεί ο κανονισμός αυτός. Αλλιώς θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος. Αντί να επεκτείνουμε την ε, απαγόρευση, να μιλήσουμε περισσότερο για την μικρή διάρκεια ανάπαυση. Για τον ταχογράφο πάντως και την ημερομηνία από την οποία θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικός. Ακούσαμε τι είπε ο εισηγητής. Λέει και η συγκήτρια ότι πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές συγχρόνως. Όταν είναι έτοιμος αυτός ευφύης ταχογράφος, τότε να δούμε. Αλλά αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα. Και αυτό πρέπει να το συμπεριλάβουμε εδώ. Για τις υπηρεσίες τώρα λεωφορείων Πούλμαν, και για δικούς κανόνες συμφωνεί και γιατί οι συνθήκες είναι διαφορετικές για αυτά τα οχήματα από ό,τι είναι για τα φορτηγά. Τώρα για να υπάρχουν εξαιρέσει σε εθνικό επίπεδο για τα οχήματα τα οποία ε, χρησιμοποιούνται στον οικοδομικό τομέα ή και για άλλες περιπτώσεις λέει η συγγήτρια ότι τα οχήματα αυτά δεν διανύουν μεγάλες αποστάσεις, οπότε δεν χρειάζονται τον εφή ταχόγραφο. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπιλμπάου. Κύριε Κιστελό, έχετε το λόγο. That's very kind of you. Thank you. Um, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βάντεκαμπ καθώς και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές για τη δουλειά που έχουν κάνει μέχρι τώρα πάνω στην έκθεση αυτή η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των κοινωνικών προτύπων των επαγγελματιών οδηγών και όσον αφορά την ασφάλειά τους και την ασφάλεια των άλλων επιβατών καθώς και των άλλων χρηστών των οδών μας. Μια παρένθεση. Απόψε στις 6 ώρα μαζί με τον κύριο Μπαχ και την κυρία Άλτετον θα συμμετάσχουμε σε στρογγυλή τράπεζα εδώ στο Κοινοβούλιο σχετικά με το χρόνο ανάπαυσης ε, των οδηγών. Ε, σας παρακαλώ λοιπόν, ε, ελάτε κι εσείς, ε, θα συμμετάσχουν και συνδικαλιστές καθώς και κάποιοι οδηγοί. Ε, προσλέπω λοιπόν στην εκδήλωση αυτή. Οι συναντήσεις των σκιωδών ε, εισηγητών ε, έγιναν με πολύ ζωντανές συζητήσεις ε, και οι συμβαστικές τροπολογίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα. Αυτή τη στιγμή εμείς οι πράσινοι είμαστε αντίθετοι με την προτινόμενη ε, τροποποίηση του περίοδου αναφορα από δύο σε τέσσερις εβδομάδες παρότι που χαιρόμαστε ότι ε, παραμένει απαράλλακτο ο μέγιστο χρόνο οδήγηση. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό να περιμένουμε από τους οδηγούς τον χρόνο ανάπαυσής τους να τον ε, περνούν στην καμπίνα του φορτηγού. Θέλουμε οι εργοδότες να ε, προβλέπουν ε, κατάλληλο κατάλημα σε ξενοδοχεία ή σε παρόμοιους χώρους ώστε να ε, αναπαυθούν καλά οι οδηγοί προτού να ξεκινήσουν την εργασία της εβδομάδας. Όσον αφορά τους ασφαλείς χώρους στάθμευσης, δεν πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο υποκαθιστά την ανάγκη των οδηγών να περνούν τον χρόνο εβδομαδίας ανάπαυσης εκτός του οχήματός τους Πολλοί θέλουν ε, να επικεντρωθούμε στην ευελιξία, αλλά διακινδυνεύουμε κινδυνεύουμε να ε, ρισκάρουμε την ασφάλεια των οδηγών, διότι η ευελιξία μπορεί να φαίνεται ότι δίνει περισσότερες επιλογές στους οδηγούς, αλλά πρέπει να προσέξουμε ε, στην πράξη αυτό να μην να μην είναι εις βάρος του χρόνου ε, ανάπαυσης. Οι οδηγοί πάντα θέλουν να πιέζουν ώστε να έχουν περισσότερες ώρες οδήγησης. Αυτό όμως είναι εις βάρος της ασφάλειάς τους και της ασφάλειας άλλων χρηστών των δρόμων. Επίσης, ε, τα ελαφρά εμπορικά οχήματα ε, χαιρόμαστε που πλέον θα συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της ε, νομοθεσίας αυτής και μάλιστα από 2,5 τόνους άνω. Ωστόσο, θέλουμε να δούμε τις παρεκκλήσεις που θα προταθούν. Η Οδηγή λεωφορείων και πούλμαν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, λαμβάνοντας υπόψη την ε, ασφάλεια ε, των επιβατών τους. Συνήθως μεταφέρουν 53, μέχρι 53 άτομα. Η κούραση στους δρόμους αποτελεί πολύ συχνά την αιτία ατυχημάτων. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι το θέμα αυτό είναι θέμα ζωής και θανάτου. Αυτή τη στιγμή είμαστε κάπως απογοητευμένοι από την κατεύθυνση που παίρνουν οι διαπραγματεύσεις πάντα. Όμως είμαστε αισιόδοξοι και προσβλέπουμε στην αυριανή συνάντηση των σκιωδών εισηγητών όπου ε, αναμφίβολα θα ξαναπροσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε λύσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τέιλορ. Κύριε Κιλάναν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί προσκεκλημένοι μας, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φαντεκάμπ για την πολύ ανοιχτή στάση του στον διάλογο μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Ευχαριστώ και τους ε, άλλους σκιώδεις εισηγητές, ε, διότι είχαμε πολύ δημιουργικές συναντήσεις και προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα και να βρούμε λύσεις για αυτά. Εμεί θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους οδηγούς να έχουν ασφαλείς ε, τόπους ανάπαυσης και τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο σπίτι τους ή να πάνε αλλού, εάν δεν θέλουν να πάνε σπίτι τους. Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια κατά τις ε, μετακινήσεις, ε, θέμα πολύ σημαντικό. Και πώς μπορούμε να πετύχουμε ευφυή επιβολή των κανόνων. Θέλουμε επίσης να έχουμε όσο γίνεται πιο χαμηλό γραφειοκρατικό άχθος στο σύστημα αυτό, αλλά και από την πλευρά των οδηγών όσον αφορά το τι θα πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους ε, στο όχημα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τι έγγραφα χρειάζεται να κουβαλούν μαζί τους ε, και στο μέλλον. Ε, τα ελαφρά φορτηγά οχήματα είναι σημαντικό θέμα και νομίζω ότι πλησιάζουμε σε μια λύση περισσότερο από ποτέ. Επίσης, όσον αφορά τις μη εμπορευματικές μεταφορές και τους οδηγούς των οποίων η κύρια ασχολία δεν είναι η οδήγηση, ο Βίμ γνωρίζει πολύ καλά ότι προσπαθήσαμε να ε, προωθήσουμε την θέση της Επιτροπής ε, Απασχόλησης ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα ελαφρά οχήματα για τη μεταφορά προϊόντων εκτός εάν χρησιμοποιούνται για το, το, τους ίδιους στόχους της εταιρείας ε, ή του οδηγού ε, ή εάν ε, η οδήγηση δεν είναι η κύρια απασχόληση του ανθρώπου που οδηγεί το όχημα. Ξέρουμε ότι το Κοινοβούλιο προσπαθεί κάθε φορά να επιβάλλει χρονικά όρια στα έγγραφα και ναι, έχουμε όριο 12 ώρων Ε, στα έγγραφα για τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης. Μαζί με τον ορισμό της οδήγησης ως ε, κύρια απασχόληση. Εγώ σύμφωνα με τον ορισμό αυτό είμαι ε, επαγγελματίας οδηγός διότι οδηγώ τουλάχιστον 12, εβδομάδες, 12 ώρες την εβδομάδα στη Φιλανδία λόγω των μεγάλων αποστάσεων. Υπάρχουν όμως άλλες χώρες με τελείως διαφορετικές ε, συνθήκες. Με πολύ πιο σύντομες διαδρομές. Αγαπητέ Βιμ, θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Μερικοί προτιμούν τις τέσσερις εβδομάδες, ε, άλλοι τρεις. Εμείς ίσως προτιμήσουμε τις δύο εβδομάδες. Όσον αφορά τους ευφυείς ταχογράφους, και το θέμα των λεωφορείων και των πούλμαν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να προωθήσει την ιδέα ότι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αναπτύξουν νέα είδη ταχογράφων, να μην χρησιμοποιείται το ίδιο είδος ταχογράφου για όλες τις επιχειρήσεις και για όλους τους τομείς. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επίτροπος και όλο το προσωπικό να προωθήσουν την ανάπτυξη πιο ευφυών ταχογράφων. Κοντεύουμε να κάνουμε τουριστικά ταξίδια στο φεγγάρι. Ε, δεν μπορεί να μην μπορούμε να αναπτύξουμε το σωστό είδος ταχογράφου. Νομίζω ότι θα με πυροβολήσει τώρα η Πρόεδρος. Καλύτερα να κλείσω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κιλένεν. Κυρία Αρνάτου, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε κύριε Σιγητή, κύριε Βαντεκάμπ, ότι έχετε κάνει πολλή δουλειά για τις συμβιβαστικέ ε, μεταξύ όλων αυτών των τροπολογιών που προτείνουν ε, αυστηρό περιορισμό του χρόνου εργασίας των οδηγών μερικές φορές και με επικίνδυνο τρόπο ε, όσον αφορά την ευελιξία αλλά τα προβλήματα τα βασικά δεν έχουν λυθεί Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι πολύ δύσκολο ή αδύνατο να βρούμε ε, σύγκληση όταν είναι τόσο αντίθετε οι απόψει, όχι μόνο λόγω πολιτικών ευαισθησιών διαφορετικών, αλλά και για οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα εθνικά που είναι πολύ διαφορετικά. Α, ιδεολογικά φτιάξαμε την Ένωση πριν να είναι αυτή εφικτή και κοινωνικά και οικονομικά. Εγώ λυπάμαι γιατί ορισμένες συμβιβαστικέ ε, δεν οδηγούν σε μεγαλύτερη προστασία των οδηγών και των συνθηκών εργασίων τους. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κάποιους από εσά, κάποιους βουλευτές που αρνούνται οποιαδήποτε πρόοδο όσον αφορά τον περιορισμό του χρόνου εργασίας, παρότι καταλαβαίνω ότι αυτό συνεπάγεται ζημίες ε, και ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις των εκάστοτε χωρών και δεν θέλω να το παρατήσουν, θέλω να σας ρωτήσω, πραγματικά ειλικρινά θα το κάνατε, αυτό το επάγγελμα υπό αυτές τις συνθήκες θα θέλατε να το κάνουν τα παιδιά σας ή τα εγγόνια σας να γίνουν οδηγοί ε, σε με τέτοιους χρόνους ε, και επιστρέφοντας στο σπίτι τους μια φορά το μήνα για να μην μιλήσουμε για τα λεφτά που κερδίζουν. Πραγματικά πρέπει να τον ερωτηθείτε. Αν η, ερώτηση, αν η απάντηση συγγνώμη, είναι αρνητική, τι να πω, δεν αλλάζει τίποτα διότι εσείς αντί να εξυπηρετείτε το γενικό ε, συμφέρον εξυπηρετεί τα επιμέρους ε, συμφέροντα. Ευχαριστούμε κυρία Αγνωτή. Κύριε Μπάχα, εκ μέρου τη Επιτροπής Απασχόλησης έχετε το λόγο γιατί είστε εισηγητής της Επιτροπής εκείνης. Ε, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης. είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Βαντεκάμπ και με τους ε, σκιώδεις εισηγητές που έχουν λάβει υπόψη τους σε πολλά από τα σημεία της νομοδότησής μας. Ε, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια θέματα. Ε, ήμασταν κατά της περισσότερης ευελιξίας, διότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν ισχύ οι ισχύοντες κανόνες. Ε, το πρόβλημα δεν είναι οι κανόνες αλλά η έλλειψη ελέγχων και οι ανεπαρκής κυρώσεις. Δεύτερο θέμα είναι η συμπερίληψη των ε, ελαφρών φορτηγών ε, στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας. Αυτό στο μέλλον θα σημάνει καταρχάς βελτίωση των ε, συνθήκων εργασίας των οδηγών ε, και βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Τρίτον, ε, απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. απαγορεύεται λοιπόν ο χρόνος ανάπαυσης στην καμπίνα του φορτηγού και μετά από τρεις εβδομάδες ε, προβλέπεται επιστροφή του οδηγού στον ε, τόπο διαμονής του ή σε άλλο τόπο της επιλογής του. Τελευταία παρατήρηση για τους ταχογράφους. Ε, οι συνάδελφοι ήδη το είπαν αυτό. Η μεταβατική περίοδος μέχρι το 2030 είναι απαράδεκτη και για μας. Πιστεύουμε ότι όσο το δυνατόν συντομότερο θα πρέπει να ε, εισαχθούν. Ε, δεν έχουμε καμία κατανόηση για τόσο μακρά ε, μεταβατική περίοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπάχα. Για δύο λεπτά λοιπόν ο καθένας ε, θα έχετε για να πείτε ό,τι έχετε να πείτε. παρακαλώ τρίστε το χρόνο. Κύριε Κόχ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Βιμ για τις ε, γενικά εξαιρετικές ε, συμβαστικές προτάσεις. Έχουμε τις ε, ισχύουσες παρεκκλήσεις, αλλά θα πρέπει τώρα να αδράξουμε την ευκαιρία ώστε να μην επιβάλλουμε επιπλέον γραφειοκρατικό άχθος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άλλωστε δεν είναι η ομάδα στόχος της νομοθεσίας αυτής. Ε, συμφωνώ με την ε, μείωση του ορίου από τους 3,5 τόνους στους 2,5 ή ακόμα και στους 2,4 ε, τόνους. Και πιστεύω ότι θα πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να υποφεληθούν από τις διατάξεις του άρθρου 3. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το όριο των 100 χιλιόμετρων από την έδρα της επιχείρησης θα πρέπει να αυξηθεί στα 150 χιλιόμετρα. Ε, άλλωστε, ε, μας ενδιαφέρει και το θέμα των ε, εργατών, για παράδειγμα, που μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους. Επίσης, δεν πιστεύουμε ότι χρειάζεται ταχογράφο κάποιο ο οποίο μεταφέρει ένα δέντρο, για παράδειγμα ένα κυπουρό μεταφέρει ένα δέντρο από την επιχείρησή του σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων. Επίσης ε, τα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων ε, δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχουν το όριο των 50 ε, χιλιόμετρων. Ας, διατηρήσουμε, ας αυξήσουμε λοιπόν το όριο στα 150 χιλιόμετρα ή υπό ιδανικές συνθήκες να το αυξήσουμε στα 200 χιλιόμετρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρικέ. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα με ικανοποιεί η εισαγωγή των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με την εξαίρεση όμως την οποία δεν καταλαβαίνω καθόλου. Όταν έχουμε ένα ταχογράφο όσους κάνουν για βιοτεχνικές δραστηριότητες μικρές αποστάσεις έχουν έναν ταχογράφο ε, επίσης δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε εξαιρέσεις εκτός αν κάνουμε χιλιομετρική εξαίρεση μετά τον έξυπνο ταχογράφο Όλοι λένε όλοι αυτοί οι κανονισμοί ε, δεν έχουν ε, ενδιαφέρον αν δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Πολύ καλό που τους εισάγουμε, καλά κάνουμε και λέμε τι πρέπει να, πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα, καλά κάνουμε και δίνουμε και μια προθεσμία. Το 2020 το υποστηρίζω εγώ. Κάτι όμως μου δημιουργεί προβληματισμούς. Αυτός ο κανονισμός ουσιαστικά είναι κοινωνικός. Γενικά από τους κοινωνικούς κανονισμούς αναμένουμε κάποια κοινωνική πρόοδο. Τώρα εξετάζοντας λεπτομερώς το κείμενο, ο χρόνος εργασίας αυξάνεται, η ανάπαυση στην καμπίνα επιτρέπεται, αντίθετα από την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά δεν είναι το δικαστήριο εκείνο που θα μας πει ποιος θα είναι ο κανονισμός. Εμείς λέμε στο δικαστήριο τι πρέπει να πει. Και τρίτον, μπορούμε να κατακαιρματίσουμε το διάλειμμα μετά μπορούμε να κάνουμε διαλύματα στις συνδυασμένες μεταφορές. Μετά η επιστροφή στο σπίτι τους. Ναι, κάποιοι οδηγοί μπορούν να μένουν στην Ισπανία δεν ξέρω εγώ και να παίζουν και εγώ όταν δουλεύω δουλεύω σπίτι μου και δεν παίζω γιουκουλέλε. οπότε αυτό που θέλω να πω μου κάνει έκπληξη ότι ένας κοινωνικός κανονισμός ουσιαστικά υπονομεύει τα κοινωνικά δικαιώματα. Ναι, ξεβελιξία, ναι, μια χαρά είναι. Αλλά είναι ανεπαρκής, εγώ πιστεύω. Λοιπόν, αφού έχετε τέτοιες αμφιβολίες, θα το εξετάσουμε. Κυρία Λουκασέσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να αναφερθώ στον ορισμό του συμβασμού, γιατί νομίζω ότι είναι μια ιδιαίτερη έννοια. Κανονικά σημαίνει κάτι το οποίο να είναι αποδεκτό από όλες τις πλευρές που συμμετέχουν στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή όλοι κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις, ε, όλοι αφήνουμε στην πάντα κάτι που μας ενδιαφέρει. Προκειμένου να επιτευχθεί ένα συμβασμό. Μόνο τότε μπορούμε να μιλήσουμε για συμβασμό. Αν ο ένα προσπαθεί να επιβάλλει στον άλλον τι επιθυμίε του, ε, τότε δεν πρόκειται για συμβιβασμό. Να το έχουμε υπόψη μα αυτό. Τώρα, όσον αφορά την έκθεση του κ. Βαντερκάμπ, χαίρομαι πολύ γιατί ήταν ανοιχτό σε κάθε είδου προτάσει, ιδέε άκουσε τα διάφορα προβλήματα που εκφράσαμε. Όσοι γνωρίζουν καλά το κλάδο, ξέρουν ότι δεν έχουμε σύστημα πιστοποίησης απόλυτο. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να δημιουργηθούν τέτοιοι σταθμοί, τέτοιοι χώροι στάθμευσης κλπ. Ο ΒΙΜ λοιπόν μιλάει για την δυνατότητα ανάπαυσης όχι μόνο σε ξενοδοχεία. Εκείνος είχε την ευκαιρία μάλιστα να ανέβει στα πιο σύγχρονα φορτηγά και είδε ότι μερικές φορές οι χώροι εκεί είναι καλύτεροι και είναι καλύτεροι ακόμα και από κάποια δωμάτια ξενοδοχείων. Υπάρχει αρκετός χώρος ώστε οι δελκέριδες να μπορούν να κοιμηθούν εκεί. Είναι μια λύση που είναι πολύ κοντά σε αυτό που μας ζητούν ήδη οι μεταφορεί και οι επιχειρήσεις τους. Όσον αφορά τον ΕΦΗ ταχογράφο, θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα έχουμε ΕΦΗ ταχογράφου που να μπορούν να λύσουν τα διάφορα προβλήματα που εντοπίζονται σχετικά με τις μεταφορές, δηλαδή μεταφορές, καμποτάζ, αποσπασμένοι κλπ. Αν ναι, Πού είναι αυτές οι επιχειρήσεις, τι μάρκα είναι αυτή η ευφύη σταχογράφη. Θα γινόταν μέσα στη χρονιά να μπορούμε να ψηφίσουμε για αυτούς τους ευφύης ταχογράφους προκειμένου να εξοπλιστούν τα φορτηγά μας με αυτούς μέσα στη χρονιά. Αν αυτό που θέλουμε είναι το 2020 οι τα ταχογράφοι να είναι μόνο στα φορτηγά, θέλω να το ξέρω, ή τους θέλουν για όλα τα οχήματα. Και έπειτα, μιλάμε για οχήματα πάνω από 3,5 τόνους. Να ξέρουμε ότι μιλάμε για ιδιαίτερα υψηλό κόστος, 1.000 ευρώ κοστίζει να εγκαταστήσει κανείς ένα νέο ταχογράφο. Δεν κατανοούν όλοι γιατί πρέπει να αναλάβουν τέτοιο κόστος 1000 ε, ευρώ για τις δραστηριότητές τους. Να τηρείτε το χρόνο μιλία σας, λέει ο Πρόεδρος, μετά θα είμαι πιο αυστηρή και θα σας κόβω το λόγο. Ε, κύριε Ντέλη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα αρχίσω με ευχαριστίες και συγχαρητήρια στον κύριο Βαντερκάμ και τους συνεργάτες του γιατί πραγματικά μας συμπεριφέρθηκαν με πάρα πολύ καλό τρόπο ήταν ανοιχτή απέναντί μα, δεν μας έκρυψαν τίποτα, οπότε χαίρομαι πολύ για αυτή την προσέγγιση. Δύο πράγματα θέλω να επαναλάβω. Για τις τέσσερις εβδομάδες ως ε, περίοδος ε, αναφοράς πρέπει να μην ξεχνάμε και την περίοδο των 180 ωρών. Δηλαδή ο χρόνος εργασίας με τον χρόνο ανάπαυσης πρέπει να σχετίζονται. Έπειτα για την μεταβατική περίοδο προκειμένου να έχουμε χώρους κατάλληλου στάθμευσης. Χρειάζεται χρόνος για να προετοιμαστούν, για να προσαρμοστεί η εθνική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις που χειρίζονται δηλαδή τους χώρους αυτούς στάθμευσης να προσαρμοστούν. Ήδη υπάρχουν κάποια εθνικά μέτρα που απαγορεύουν ε, στους ε, φορτηγούς να κοιμούνται μέσα στα φορτηγά τους αν δεν υπάρχουν ε, οι κατάλληλες συνθήκε. Αυτό όμως είναι υποκριτικό γιατί πώς θα το ελέγξουν. Είχα κάποιους Ρουμάνους οι οποίοι τιμωρήθηκαν στη Γαλλία και το Βέλγιο γιατί δεν κοιμήθηκαν στο ξενοδοχείο τους, δεν κοιμήθηκαν μέσα στο φορτηγό τους, έξω από αυτό, αλλά τους τιμώρησαν παρόλα αυτά γιατί δεν πήγαν στο ξενοδοχείο. Μα τότε καταπιέστη η ελευθερία προσφοράς υπηρεσιών. Είναι θέμα ευρωπαϊκό η νομική βεβαιότητα για κανόνες και με κανόνες οι οποίοι να είναι ρεαλιστικοί. Οπότε θα ήθελα να υπάρχει νομική προστασία στις επιχειρήσεις και στους οδηγούς κατά τέτοιων μέτρων που τους τιμωρούν. Το έχω πει πολλές φορές μέχρι τώρα. Χρειαζόμαστε ρεαλιστικά μέτρα, ε, βιώσιμες λύσεις και ελπίζω να τα καταφέρουμε στο τέλος αλλά πριν τις 4 Ιουνίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντελή. Η κυρία Κρατσφάτερ έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, πρέπει να βρούμε εφικτές λύσεις, αλλά ποιος είναι ο στόχος αυτών των νέων διατάξεων. Η βελτίωση είναι ο στόχος μας ε, των συνθήκων εργασίας, της ασφάλειας ε, στις οδικές μεταφορές και θέμη το ανταγωνισμό ανάμεσα στους οδηγούς όλων των κρατών μελών. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Νομίζω σε αυτό συμφωνούμε. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε ε, ανάλογα βήματα. Η ευελιξία στον χρόνο εργασία ακούγεται πολύ ωραία, αλλά συνήθω είναι ει βάρο των συνθήκων εργασία των οδηγών και τη ασφάλεια στις οδικές μετακινήσεις και θα πρέπει ε, και σε αυτό να εστιάσουμε. Όσον αφορά του ευφυεί ταχογράφου, εγώ βρίσκω περίεργο το 2018 ε, να ε, θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι τόσο δύσκολο. Θα πρέπει να είναι σχετικά εύκολο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τρομερή τεχνογνωσία Το θέμα είναι πώς θα ελέγξουμε την κατάσταση αν δεν έχουμε αυτούς τους ταχογράφους. Επίσης, ε, η διανυκτέρευση στην καμπίνα του οδηγού. Νομίζω ότι ο ε, εκτενή χρόνος εργασίας δεν θα πρέπει να περνιέται στην καμπίνα του οδηγού. Δεν θέλουμε νομάδες ε, στους δρόμους της Ευρώπης. Και εάν θέλουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των οδηγών, θα πρέπει να τους προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες εργασίας, ε, κάτι το οποίο δεν συνάδει με το χρόνο ανάπαυσης ε, στην καμπίνα του οδηγού. Τους ε, οδηγούς φορτηγών θέλουμε να τους διατηρήσουμε στο επίκεντρο, θέλουμε να πετύχουμε καλές συνθήκες εργασίας και κάτι τέτοιο θα το πετύχουμε μόνο με καλές συμβαστικές προτάσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κομπάσεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω πρώτα απ' όλα μία ερώτηση. Ποιε συμβιβαστικέ τροπολογίες συζητάμε σήμερα, διότι από ό,τι κατάλαβα συζητούσαμε τις συμβιβαστικέ που θα ψηφιστούν αύριο το πρωί. Εγώ δεν έχω λάβει τις συμβιβαστικέ τροπολογίες και εγώ πρώτη φορά βλέπω να συζητάμε κάτι για το οποίο δεν έχουμε κανένα χαρτί, δεν το έχουμε λάβει. Κάποιοι συναδελφοί λένε τέσσερι εβδομάδε, άλλοι λένε δύο εβδομάδε. Εγώ να προτείνω δεκάξι. Όταν συζητάμε συμβιβαστικέ τροπολογίε, πρέπει να μα τι δίνετε στα μέλη τη Επιτροπή για να μπορούμε να τι συζητήσουμε κανονικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαντεκάμπ και να τον συγχαρώ που αισθάνεται καλά. Αλλά ξέρετε, τα συναισθήματα στη δική μου χώρα είναι λίγο διαφορετικά. Αύριο η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Μακρόν θα βρίσκονται στη Σόφια και εκεί θα δουν με τα ίδια τους τα μάτια μια τεράστια διαδήλωση διαμαρτυρίας των οδηγών φορτηγών. Σε συγχαίρω που σας νοιάζουν τόσο πολύ οι βουλγαρικές ε, οικογένειες. Μόνο οι εκκλησίες έχουν δείξει τέτοια συμπόνια. Ίσως θα μπορούσατε να θέσετε υποψηφιότητες στη Βουλγαρία. Θα λάβετε την υποστήριξη εκεί πολλών ε, οικογενειών. γιατί να μην απαιτείται να έχουν επιστρέψει οι οδηγοί στα σπίτια τους μέχρι, μέχρι συγκεκριμένες ώρες. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω τους εισηγητές, ε, όταν αναφέρουν τις πολιτικές ομάδες, θα θέλαμε να πούν κατά πόσο μιλούν εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων των κρατών μελών στα οποία ανήκουν και τα οποία τους έχουν εκλέξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ερτούγκ, έχουμε προσκεκλημένο στην Επιτροπή μας. Από το Ίδρυμα Ρομπέρτ Σούμαν. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλώς ορίσατε. Να τους χειροκροτήσουμε. Και συνεχίζουμε τις αξίες μας για τη δεσμεμέτρα για την κινητικότητα και ο τελευταίος ομιλητής είστε εσείς κύριε Ερτούγκ. Για λιγότερο από δύο λεπτά έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Φάντε Κάμπ για την πρότασή του αυτή. Πράγματι, είναι δύσκολο θέμα, διότι τα τρία νομοθετικά αυτά θέματα σχετίζονται μεταξύ τους και υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από χώρες ε, της Κεντρικής ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της περιφέρειας και είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσουμε τα διάφορα συμφέροντα σε μια ενιαία πρόταση. μιλούν διάφοροι, αλλά κάποιος ε, που τα ακούει αυτά απ' έξω είναι πολύ δύσκολο να κρίνει ε, ε, εκ μέρους ποιου τα λέει κανείς αυτά. Όσον αφορά τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία υπέρ του να μην περνιέται ο χρόνος ανάπαυσης μέσα στην καμπίνα του οδηγού. Και επίσης, ο οδηγός μετά από συγκεκριμένο αριθμό εβδομάδων θα πρέπει να επανέρχεται στην χώρα διαμονής του ώστε να περάσει το χρόνο ανάπαυσής του στο, στον κοινωνικό του περίγυρο το μετά από πόσε εβδομάδε θα πρέπει να γίνεται αυτό, αυτό θα είναι αντικείμενο πολιτική συζήτηση. Και εντό τη δική μου πολιτική ομάδα υπάρχουν προτάσει από δύο έω, τι να σα πω, οχτώ εβδομάδε. Η πλειοψηφία τη σοσιαλιστική ομάδα είναι υπέρ δύο, το πολύ τριών εβδομάδων. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν οδηγώ από Δευτέρα μέχρι Σάββατο με περιορισμένο χρόνο ανάπαυσης και μετά πρέπει να ξαναοδηγήσω Δευτέρα με Παρασκευή. Νομίζω ότι συσσωρεύεται ο χρόνος ανάπαυσης των δύο δηλαδή εβδομάδων, δηλαδή μισή μέρες τις οποίες πρέπει να περάσω στο χρόνο διαμονής μου. Ε, το λέω αυτό έτσι ξεκάθαρα, διότι συγχωρήστε με, αλλά Ε, ε, ακόμα και εμεί ε, μετά από ένα Στρασβούργο για παράδειγμα, Πέμπτη, ήδη βιαζόμαστε όλοι να φτάσουμε σπίτι μας. Γιατί να είναι διαφορετικά τα πράγματα για τους οδηγού φορτηγών. Εάν λοιπόν έχουν εργαστεί πέντε μέρες και μετά άλλες έξι, έντεκα μέρες λείπουν από το σπίτι τους. Οδηγώντας και μπορεί να λένε κάποιοι ότι οι χώρες της περιφέρειας ε, αντιμετωπίζουν διαφορετική κατάσταση αλλά θα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε νομικό πλαίσιο και δεν επιτρέπεται να νομοθετήσουμε ώστε να επιτρέπεται να γίνει κάτι τέτοιο. Και τελευταία μου πρόταση με τα αποτελέσματα. Είδαμε ποια είναι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, είναι μια θέση πολύ κοντά στη θέση των ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας. Ε, παρακαλώ λοιπόν όλους να προσεγγίσουν το θέμα αυτό με λογική. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Γιατί κοιτάτε έτσι κύριε Βαντεκάμπ, θα σας δώσω το λόγο. Μετά θέλω να ακούσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Λιζόα, έχετε το λόγο για αυτό το πρώτο σημείο που αφορά τους χρόνους ανάπαυσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές. Βλέπουμε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα φιλόδοξη έκθεση προκειμένου να αρχίσει να ισχύει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία με τα ψηφιακά δεδομένα. Χαιρόμαστε γι' αυτό και ξέρουμε ότι και ο κύριος Βαντερκάμπ είναι πάρα πολύ λογικός άνθρωπος, οπότε η λύση που προτείνει είναι αναλογική. Και συνεπώς πολύ χαιρόμαστε γι' αυτή, γιατί δεν θα επιβάλλει μεγάλο επιπλέον κόστος ούτε στις εθνικές δικήσεις, ούτε στους επιχειρηματίες, προκειμένου να επιβληθούν τα νέα μέτρα. Οπότε, πολύ χαίρομαι για τις προτάσεις σας που περιλαμβάνουν λογικές λύσεις. Σύντομα, θέλω να αναφερθώ σε τρία σημεία. Πρώτον, για τους χώρους στάθμευσης που αναφέρεται. Ο έλεγχος και η καλύτερη χρήση επίσης των ταχογράφων με απασχολεί. Λοιπόν, για το πρώτο, για του χώρου στάθμευση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το συζητήσαμε, όπως ξέρετε, στο Συμβούλιο, όπου διάφορες χώρες μέλη έχουν εγκρίνει μέτρα ε, αποτροπής να περνάνε τα Σαββατοκύριακά τους στα φορτηγά τους, η Γερμανία, το Βέλιο, η Γαλλία για παράδειγμα αλλά αναρωτιόμαστε, βελτιώνονται οι συνθήκε εργασία εξαιτία τη απαγόρευση αυτή. Η απάντηση είναι όχι. Άρα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση. Η ανάπτυξη προφανώ τέτοιων ασφαλών και αναπαυτικών χώρων στάθμευσης για τα φορτηγά. Παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις και έχουμε υπόψη μας την τροπολογία Βαντερκάμπ όπου λέει ότι το Σαββατοκύριακο να μπορεί να ε, το περνάει στο φορτηγό του εφόσον είναι σταθμευμένο σε έναν κατάλληλο χώρο. Λοιπόν, μπορούμε να συμφωνήσουμε και το έχουμε πει αυτό και νωρίτερα. Ο εισηγητής επίσης θεωρεί ότι η ανάπαυση ε, στα φορτηγά πρέπει να απαγορεύεται και για την, ε, το μειωμένο χρόνο ανάπαυσης. Ο οδηγός λέγαμε πριν ότι μπορούσε να μένει στο φορτηγό του για τον μειωμένο χώρο χρόνο ανάπαυσης. Και αυτό υποστηρίζουμε και τώρα. Για τα δεδομένα. Σίγουρα τα διάφορα στοιχεία και τα δεδομένα θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ να ελέγχουμε την ε, εφαρμογή των μέτρων αυτών. Ευχαριστώ και τον κύριο Ερτούκ και την κυρία Κίλωνεν Και πρέπει πράγματι ό,τι μέσα έχουμε ήδη στη διάθεσή μας για τη συλλογή στοιχείων να τα χρησιμοποιήσουμε στο επακρόν για να μπορούμε να βοηθηθούμε χωρίς επιπλέον κόστος από πλευράς των εθνικών δικήσεων. Τέλος για τον ταχογράφο. Σημειώνω τις τροπολογίες σας που στηρίζουν διάφοροι ευρωβουλευτές όσον αφορά τους κοινωνικούς κανόνες και τον ταχογράφο στα ελαφρά εμπορικά οχήματα. Η Επιτροπή, όπως ξέρετε, πρότεινε να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Δηλαδή, ε, μόνο για την πρόσβαση στο επάγγελμα, όταν πρόκειται για τα ελαφρά οχήματα. Για το retrofit σημειώνουμε τις εξελίξεις. Είναι αλήθεια ότι το 2018 δεν φαίνεται να είναι λογικό οχήματα σε διεθνείς μεταφορές να εξακολουθούν να κυκλοφορούν με αναλογικούς ε, ταχογράφους. Εξού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ημερομηνίες για το retrofit προκειμένου να εξοπλιστούν με φύση ταχογράφους τα φορτηγά το 2026. Και ολοκληρώνω απαντώντας κάπως σύντομα για το ζήτημα αυτό των αρχιών ταχογράφων ακριβώς. Θα λύσουν όλα τα προβλήματα. Κατά πάσα πιθανότητα όχι, δεν θα λύσουν όλα τα προβλήματα. Θα βελτιώσουν όμως την εφαρμογή των μέτρων δεδομένου ότι θα γνωρίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την ακριβή τοποθεσία του φορτηγού. Ελέγχονται λοιπόν αυτοί οι ευφύς ταχογράφοι και θα εγκατασταθούν από τα μέσα του 2019 στα νέα φορτηγά. Είναι κάτι που δέχονται διάφορες εταιρείες, η Sonwich και η Continental, για παράδειγμα. Αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη δέσμη αυτή μέτρων. Ευχαριστούμε κύριε Λιζουά. Είπατε χώρη στάθμευσης ασφαλής και αναπαυτική. Τι σημαίνει όμως αυτό μπορείτε να μας πείτε. Δεν μπορούμε να πούμε απλώς ένα ξενοδοχείο, ένα μοτέλ, ένας χώρος που να μπορεί κάποιος να Γιατί τι σημαίνει πάρκινγκ αναπαυτικό. Καταλαβαίνετε. Αν πρέπει μετά να περάσουμε από κατεξουσιοδότηση πράξης θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λυπάμαι. Ένα πάρκινγκ ασφαλέ και αναπαυτικό δεν σημαίνει τίποτα. Κάποιο μπορεί να μου το εξηγήσει τι σημαίνει. Α, ο κύριο ε, Βαντεκάμπ μπορεί να μου το εξηγήσει πολύ ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά πρέπει να σας πω ότι πάρα πολύ ωραία πάντα πράγματα. Η πρότασή μου μπορεί βεβαίως να βελτιωθεί παρετέρω. 16 εβδομάδες λένε κάποιοι μακριά από το σπίτι τους οι οδηγοί από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά λένε 4 εβδομάδες και έχω και τον συνάδελφο Ερτούκ που λέει 2 εβδομάδες. Οπότε εγώ είμαι βασιλιάς των δρόμων. Τι να σας πω, πώς να καταλήξω σε συμβιβασμό. Γι' αυτό είπα ανάμεσα στις τρεις και τις τέσσερις εβδομάδες εκτός έδρας. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Εδώ θα μπορούσαμε να μιλάμε επάπειρο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην καταλήξει πουθενά. Ή να βάλουμε τη λογική μας να δουλέψει και να καταλήξουμε σε λογικούς συμβασμούς. Η επιλογή είναι δική σας. Η δικιά μου η πρόταση είναι ξεκάθαρη. Αύριο άλλη μια φορά θα μιλήσουμε με τους σκιώδεις και μετά θα καταλήξω σε μια συμβαστική πρόταση. Και όλοι γνωρίζουν, εκτός από τον κύριο Πέτρο Κομπατσέφ, τον συμβασμό, άρα δικό του θέμα είναι. Τι να κάνω. Και για τις άλλες προτάσεις μπορούμε να συζητήσουμε διάφορους ε, άτυπους συμβασμούς, αλλά δεν θέλουμε να φέρουμε πανικό στην Ευρώπη. Τώρα για το περίφημο going home, πώς επιστρέφει κανείς σπίτι του, στην έδρα του. Δεν φαίνεται να το καταλαβαίνουν όλοι, δεν θέλουν. House is house. Το να γυρνάει κανείς σπίτι του σημαίνει ότι γυρνάει σπίτι του. Αν πω ότι δεν θέλω να πάω σπίτι μου, αλλά θα πάω στην Αραγώνα, στην ε, παράνομη φιλενάδα μου, ε, αυτό δεν είναι σπίτι. Η επιχείρηση δεν θα σου πληρώσει εισιτήριο για να πας στην Ταραγώνα. Θα σου πληρώσει εισιτήριο για να γυρίσεις στη Σόφια, εφόσον στη Σόφια μένεις. Χώρος κατοικίας είναι ο χώρος κατοικίας. Αν συνονιθείς ότι δεν θέλεις να πας στο σπίτι σου αλλά στην παράνομη φίλη σου στην Ταραγώνα, τότε μπορείς αυτό να το συμφωνήσεις με τον εργοδότη σου. Αλλά δεν πρέπει εμείς να καθόμαστε τώρα να συζητάμε και να λέμε ότι δεν είναι σαφές το ποιο είναι το σπίτι του καθενός. Ε, είτε πρόκειται για ομοφιλόφιλους, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο που δεν θέλουν να πάνε στο ένα μέρος, αλλά θέλουν να πάνε στο άλλο. Εμείς αναγνωρίζουμε το χώρο κατοικίας. Τελείωσε. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Σπίτι. Για επιστρέψτε στο θέμα, κύριε Φαντέκο, και μην ε, εδώ πέρα σπάτε καρδιές. Αν κάποιο εδώ λέει ότι δεν το καταλαβαίνει, δεν θέλει να το καταλάβει αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για την ανάπαυση μέσα στο φορτηγό. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο μεγάλος χρόνος ανάπαυσης, το μεγάλο Σαββατοκύριακο ας πούμε, λέμε ότι θα μπορού, ότι θα πρέπει να μην γίνεται μέσα στο φορτηγό. Αλλά ο μειωμένο χρόνο ανάπαυση που είναι 24 ώρε, αυτό θα μπορούσε. Για τις 3-4 εβδομάδες σας είπα τη γνώμη μου. Για το ταχογράφο, εντάξει θα πονέσει. Αλλά συμφωνώ με τον συνάδελφο των σοσιαλιστών από την Αυστρία. Τεχνολογικά πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε αυτούς τους ταχογράφους. Δεν θα μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε ταχογράφο στα φορτίγα αν δεν υπάρχει βούληση. «800 ευρώ στοιχίζει ένα ταχογράφος. Αν μια επιχείρηση είναι διατεθειμένη να εξοδεύει 50.000 για ένα σωρό άλλων εξοπλισμού, δεν είναι τίποτα τα 800 ευρώ. Τώρα για το θέμα του ύπνου. Εσείς μπορείτε να πάτε σε ένα ε, κακό ξενοδοχείο και μαζί με άλλες ε, τρεις ε, οδηγούς φορτηγών θα ξυπνήσετε με το, την πρώτη που θα μπει στο χώρο, δεν θα έχετε την ησυχία σας δηλαδή. Εγώ μπορεί να κοιμηθώ μέσα στο φορτηγό μου και να έχω την ησυχία μου και να μπορέσω να κοιμηθώ πολύ καλύτερα από εσά. Η αγορά περιμένει για τους ταχογράφους συγκεκριμένους κανόνες άπαξ και καταλήξουμε σε τέτοιους καθαρούς κανόνες θα ακολουθήσει και η αγορά. Αν η γαλλική κυβέρνηση δεν θέλει ε, οδηγούς φορτηγών από την Ανατολική Ευρώπη, ε, θα γκρινιάζει για το χώρο στάθμευσης. Δεν είναι ξεκάθαρη κι αυτή. Πρέπει να μιλάμε για έναν κατάλληλο χώρο και για τους Γάλλους οδηγούς φορτηγών που βρίσκονται στο Ταλίν, για παράδειγμα, να ισχύει για όλους. Ευχαριστώ κύριε Βαντεκάμπα αλλά δεν απαντήσετε στην ερώτησή μου. Τι θα πει ασφαλής χώρος στάθμευσης και άνετος. Εσείς επ' αυτού είπατε ξενοδοχείο. Δηλαδή μιλάμε για ξενοδοχείο, οπότε τι γίνεται. Το ζήτημα ξενοδοχείο σημαίνει ξενοδοχείο. Τελεία και παύλα. Εντάξει, θα το ξανασυζητήσουμε αργότερα μαζί. Μην το ανοίγουμε το θέμα τώρα. Πάμε στη δεύτερη συζήτηση. Αφορά την οδηγία των Απασπασμένων εργαζομένων. Η έκθεση της κυρίας Μέρια Κιλάναν. Να υπενθυμίσω ότι για την έκθεση για τους χρόνους ανάπαυσης του κυρίου Βαντεκάμπ θα ψηφίσουμε 4 Ιουνίου στις 4. Συνεχίζουμε. Έκθεση της κυρίας Κιλόνεν. Έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chair. Dear ladies. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες και κύριοι. Τι να σας πω για τα εμπόδια, για τα φορτηγά και αν τα κρεβάτια είναι καλά, εξαρτάται το αν είναι παλιά ή καινούργια. Αν είναι καινούργια είναι καλύτερα από τα ξενοδοχεία. Ε. τα έχω δοκιμάσει, μην νομίζετε. Λοιπόν, ας πάμε στο Lex Specialis, ε, απόσπαση εργαζομένων. Αφορά ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για έγγραφα, έξυπνη ε, εφαρμογή, έξυπνους ταχογράφους. Σχετίζεται με το καποτάζ περιλαμβάνει ιδέες για μια πλατφόρμα εμπιστοσύνης και για μια ε, ε, ε, και για την ανάληψη ευθυνών στον τομέα των μεταφορών. Αλλά αυτά τα θέματα είναι ίσονο σημασία αυτή τη στιγμή. Η απόσπαση των εργαζομένων είναι το μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή και αφορά τις διεθνείς μεταφορές. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα? που προσπαθούμε να επιλύσουμε με όλα αυτά. Ποιο είναι το κεντρικό ζήτημα που πρέπει να ε, στο οποίο πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ότι πρέπει να δώσουμε τέρμα στην στιγμή εκμετάλλευση των οδηγών που οδηγεί στο να μένουν μακριά από τα σπίτια τους και από ανθρώπους με οικογένειες, σπίτια και φίλους ε, τους μετατρέπει σε νομάδες. Γιατί ποτέ δεν επιστρέφουν σπίτι τους. Αυτό προσπαθούμε να επιλύσουμε εδώ. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια πιο υγιή, πιο ανταγωνιστική κατάσταση για όλες τις οδικές μεταφορές. Όλο τον τομέα. Κάποιοι άνθρωποι είναι απολύτως ικανοποιημένοι με την υπάρχουσα νομοθεσία, αλλά να ρωτηθείτε το εξή. Μας έχει κάνει πράγματι χαρούμενου, όλο αυτό. Όχι. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ σήμερα και μελετάμε τον κανονισμό για την απόσπαση εργαζομένων. Ξέρουμε ότι η Επιτροπή ΕΜΠΛ για αυτόν τον τομέα υψηλής κινητικότητας ε, προτείνει διάφορα ε, απόσπαση από την ημέρα αριθμό 1 ότι οποιοδήποτε δηλαδή περνάει τα σύνορα βρίσκεται σε κατάσταση απόσπασης. Καταλαβαίνουμε τι θα πει αυτό. Το θέλουμε. Καταλαβαίνετε τι κάνουμε. Αν περάσει αυτή η πρόταση. Εμένα μου έχουν πει ότι δεν χρειάζεται να το σκεφτόμαστε. Ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να ρυθμίζουμε, να νομοθετούμε, αυτή είναι η δουλειά μας. Ο κόσμος στον πραγματικό κόστος θα προσαρμοστεί στα δικά μας. Ε, λοιπόν, ε, σε έναν ιδανικό κόσμο μπορεί και να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά στην πραγματικότητα όχι. Αν ήταν να συμβεί κάτι τέτοιο, τότε γιατί έχουμε τόσες πολλές μηνύσεις στα δικαστήρια, τόσες πολλές προσφυγές. Οπότε ας εστιαστούμε στο πραγματικό πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα, πιστεύω, δεν αφορά τις εταιρείε και τους οδηγούς που παραδίδουν φορτία από τη μια χώρα στην άλλη και που ενδεχομένως ε, πραγματοποιούν και καμποτάζ καθοδόν ώστε να μην οδηγούν άδεια φορτηγά διότι οι περισσότεροι από αυτούς επιστρέφουν σπίτια τους. Το ταξίδι μπορεί να διαρκέσει μια εβδομάδα, μπορεί να διαρκέσει παραπάνω. Όπως και να έχει το πράγμα, κάποια στιγμή πηγαίνουν στο σπίτι τους. Το πρόβλημα είναι, όπως έχω ήδη πει, οι εταιρείε που εκμεταλλεύονται τους οδηγούς, τους στέλνουν σε ταξίδια και δεν τους επιτρέπουν να επιστρέψουν σπίτια τους. Το κάνουν αυτό ώστε να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Και έτσι πληρώνει το τίμημα όλο ο τομέας. Γιατί εμείς ως νομοθέτες μας αρέσει να έχουμε λύσεις ε, προσαρμοσμένες για όλες τις περιπτώσεις. Και τώρα προσπαθούμε να έχουμε ένα κανονισμό με μια ομαδική ε, κύρωση διότι υπάρχει ένα σάπιο μήλο μέσα σε ένα ολοκληρό καλάθι με καλά μήλα οπότε εγώ αυτό το ερώτημα έθεσα στον εαυτό μου και ελπίζω να κάνετε το ίδιο κι εσείς σύμφωνα με την ομοθεσία που μελετάμε, οποιοδήποτε παραβιάζει τους κανόνες, ποιος είναι αυτός, πώς θα τιμωρείται, πώς, ε, ποιος έχει το βάρος της απόδειξης και πώς θα πραγματοποιείται η απόδειξη. Ποια θα είναι η κύρωση, θα είναι αναγκαία η κύρωση, πώς θα γίνεται, πώς θα επιβάλλω, πώς θα εφαρμόζω την νομοθεσία και πώς θα την παρακολουθώ. Και τι γίνεται με τους οδηγούς και τους ε, εργοδότες τους, τις εταιρείες και τις αρχές επιβολής του νόμου. Πώς θα μπορούσαν όλοι αυτοί να το εφαρμόζουν αυτό στην καθημερινότητα, στην καθημερινή ζωή. Και κάτι άλλο που με έχει απασχολήσει πολύ. Έχει νόημα αυτή η ιδέα. Θέλουμε πραγματικά οι οδηγοί Πούλμαν που οδηγούν μια ομάδα τουριστών, ένα γκρουπ τουριστών να, να πάνε να κάνουν σκι στη Γαλλία από τη Γερμανία και παίρνουν την ίδια ομάδα για να την, το, ίδιο γκρουπ για να το επιστρέψουν πίσω αυτή είναι αποσπασμένη ή ένας οδηγός από την Ιταλία που παραδίδει ζαμπόν πάρμας ε, στην Γαλλία και επιστρέφοντας πάει η Τσεχία και η Αυστρία για να πάρει ένα άλλο φορτίο για την Ιταλία διότι είναι διαφορετικοί οι περιβαλλοντικοί κανόνες αλλά λένε ότι δεν πρέπει να οδηγάς με άδεια φορτηγά. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν κανόνες απόσπασης σε αυτές τις δύο περιπτώσεις με όλες αυτές τις διοικητικές απαιτήσει που υπάρχουν που σχετίζονται με την απόσπαση. Δεν είναι απλά ένας νόμος όλο αυτό. Συνεπάγεται σοβαρά πράγματα στην καθημερινότητα δεν θα, ήταν πιο λογικό να εφαρμόζεται όταν έχουμε ανθρώπους που περνούν μήνες να οδηγούν με φορτία από τη μια χώρα στην άλλη χωρίς τη δυνατότητα να επιστρέψουν σπίτια τους. Σε κάθε περίπτωση ο κανόνας ε, απόσπασης από μόνος του, ο κανονισμός απόσπασης δεν αποτελεί λύση για αυτά τα προβλήματα για να προστατεύσουμε τον τομέα και τους οδηγούς χρειαζόμαστε μια νομοθεσία καμποτάς για χρόνους οδήγησης ε, ανάπαυσης ε, για τις εταιρείε γραμματοκιβώτια, το καμποτάζ, όλα αυτά απαιτούνται σε καλή συνεργασία μεταξύ τους και μεταξύ μας. Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας ολόκληρη την εικόνα και όχι μόνο να λαμβάνουμε υπόψη δύο επιμέρους περιπτώσεις. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί ώστε να δώσουμε τέλος στην απληστία που βρίσκεται μέσα σε όλους μας και που ρίχνει τόσο πολύ τις τιμές των μεταφορών που ο κόσμος δεν αμείβεται σωστά για την πολύ σημαντική δουλειά που κάνει χωρίς κανένα σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Και τώρα ερχόμαστε στο μείζον ερώτημα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε αυτό τον οίκο, σε, μεταξύ μας ε, ε, που είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας ψήφισαν και μας εμπιστεύτηκαν οι ψηφοφόροι μας, οι πολίτες, ε, οι λαοί των χωρών μας θα πάρουμε τον εύκολο δρόμο ή τον δύσκολο δρόμο αυτόν που είναι γεμάτος λακκούβες. Θα συνεργαστούμε για να καταλήξουμε να έχουμε έναν έξυπνο κανονισμό ώστε να καλύψουμε τα παραθυράκια στον τομέα των μεταφορών. Αυτή τη στιγμή το μόνο που ακούω είναι δύο φωνές. Όχι ειδικό νόμο που σημαίνει ε, θέση της Επιτροπής ΕΜΠΛ όλα από την ημέρα υπαριθμών 1 όπως και σε άλλους τομείς. Χρειαζόμαστε όμως έξυπνη επιβολή του νόμου, χαμηλή γραφειοκρατία, όχι μόνο για τους οδηγούς, και για τους οδηγούς, όχι μόνο για τις εταιρείε. Και έτσι θα λυθούν τα προβλήματα. Τα προβλήματα λύνονται όχι μόνο θεωρητικά επί χάρτου. Τι να κάνουμε, να λέμε απλά τι ωραία νομοθεσία είναι αυτή που έχουμε. Θέλουμε λύση των προβλημάτων στην πραγματική ζωή. Ή αλλιώ έχουμε τη δεύτερη οδό που μα λέει να εξαιρέσουμε τι διεθνεί ε, μεταφορέ ε, από την απόσπαση. Στην πραγματικότητα, καμία από αυτέ τι λύσει δεν είναι συμβιβαστική αλλά είναι τόσο εύκολο να λέμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα. Χρειαζόμαστε έναν ευέλικτο κανονισμό για το εισοδικές μεταφορές. Να έχουμε μια νομοθεσία που να μπορεί πραγματικά να εφαρμοστεί και όχι να μας οδηγεί στα δικαστήρια όπως γίνεται σήμερα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Αυτά να γνωρίζω οι εκλογές έπονται εγώ το κάνω εδώ και 22 χρόνια. Ξέρετε, πάντα έρχονται εκλογέ. Θα αφήσουμε αυτό το ζήτημα και το φόβο να μας οδηγούν στη λήψη αποφάσεων ή τώρα ή ποτέ. Δεν μπορούμε να έχουμε νίκη για μερικούς και ήττα για όλους. Όλοι θα πρέπει να δείξουν ευελιξία και να βρούμε κάποια μέση λύση, ε, κάποια εφαρμόσιμη λύση, ώστε να δημιουργήσουμε πραγματικά δίκαιο ανταγωνισμό και να αναχαιτήσουμε την απληστία και την κατάχρηση των οδηγών. Έτσι, η κυρία Κιλόνεν είναι έτοιμη για ειρήνη μετά από σκληρή δουλειά, ένα πραγματικό συμβιβασμό, ώστε να λύσουμε τα προβλήματα με λογικό, ε, ισορροπημένο τρόπο. Είμαι έτοιμη. Είστε εσείς, αγαπητοί μου συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κίλεναν, συνεχίζουμε. Ο κύριος Τέλη. Τρία λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ ε, ανοιχτή προσέγγιση της στο δύσκολο και ευαίσθητο αυτό θέμα. Χαίρομαι πολύ που κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των σκιωδών εισηγητών μπορέσαμε να ξεκινήσουμε με πολύ καλή κατεύθυνση, διότι η πλειοψηφία επέλεξε τη συμβαστική πρόταση που αποκλεί τις διεθνείς μεταφορές από τους κανόνες για την απόσταση απόσπαση. Συγγνώμη. Ε, ήταν πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα, αλλά πρέπει να ρυθμίσουμε και κάποιες λεπτομέρειες και θα ήθελα να αναφέρω κάποιες ανησυχίες που συνδέονται με τις ε, τελευταίες, τις πιο πρόσφατες συμβαστικές προτάσεις. Καταρχάς όσον αφορά την επιστροφή στον τόπο διαμονής του οδηγού και του οχήματος. Πέρα από το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό το μέτρο αυτό και το ότι, τα ότι οι δύο εβδομάδες που προτείνονται είναι πολύ ε, σύντομο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ να δεχτώ να πρέπει να επιστρέψει και το όχημα, διότι αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα ε, κοινωνικά δικαιώματα των οδηγών ε, έχει καλός, αλλά δεν βλέπω τι ρόλο παίζει το όχημα εδώ. Η επιστροφή του οχήματος δηλαδή στη βάση του οδηγού. Ήδη έχουμε ε, επιχειρηματικά λειτουργικά μοντέλα που στόχο έχουν ε, την ελαχιστοποίηση των ε, διαδρομών από κενά οχήματα. Θα πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι όσον αφορά τις περιφερειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύσκολη η επιστροφή για τον οδηγό, αλλά το να πρέπει να μεταφέρει και το φορτηγό, αυτό είναι ακόμα πιο πολύπλοκο. Δεύτερη παρατήρηση. Οι συνδυασμένες μεταφορές και το οδικό σκέλος. Σύμφωνα με την συμβαστική πρόταση θα πρέπει να καλύπτουν ε, να καλύπτονται από τους ε, κανόνες περί απόσπασης. Η πολυτροπικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για την ε, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και μείωση των εκπομπών. Οι οδικές διαδρομές όμως θα είναι μικρής απόστασης και γι' αυτό νομίζω ότι θα είναι μάλλον αντιπαραγωγική η πρόταση αυτή. Επίσης ήταν σαφές ήδη από την αρχή ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε επιπλέον άχθος στους οδηγούς όσον αφορά δηλαδή ε, την τεκμηρίωση που θα πρέπει να κρατούν μαζί τους. Θα πρέπει ο οικονομικός φορέας να φέρει το βάρος αυτό. Δυστυχώς όμως ε, στο πιο πρόσφατο κείμενο βλέπω οπισθοδρόμηση διότι επανεμφανίζονται εδώ οι οδηγοί. Ενώ θυμάμαι σαφώς ότι είχαν υποβληθεί συγκεκριμένες τροπολογίες της εισηγήτριας που πήγαιναν προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή οι οδηγοί να απαλλάσσονται από την ευθύνη αυτή. Τέταρτον, ε, το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Μισθοδοσίας που προβλέπεται σε συμβαστική πρόταση να εισάγεται ε, με, εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι εδώ θέτουμε επικίνδυνο προηγούμενο. Δεν υπάρχει αυτό σε καμία άλλη πρόταση, είτε μιλάμε για απόσπαση είτε όχι. Αυτό επίσης επαρεμβαίνει στην κυριαρχία των κρατών μελών. Και τελευταία παρατήρηση. Υπάρχει σαφή σε σχέση ανάμεσα σε όλα αυτά τα θέματα και Βλέπω ότι το λέξη specialis στην περίπτωση αυτή εξαρτάται από την νομοθεσία περί εντομεταφορών. Ε, όλοι μιλούν για τους ευφυείς ταχογράφους ως την καλύτερη λύση, αλλά ε, τίθενται πολλά θέματα, το κόστος για την επιχείρηση κλπ. Ίσως ε, θα έπρεπε να επανέλθουμε σε μια πιο απλή παραδοσιακή μέθοδο, όπως οι απλές δηλώσεις ε, εντομεταφορών για να βοηθήσουμε έτσι την καλύτερη επιβολή των κανόνων. Θα κλείσω εδώ και προσλέπω στη συνέχιση των, της συνεργασίας με τον εισηγητή τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιάλα Σέντερ, καλημέρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Για τον κύριο Φαντερκάμπ εγώ ήθελα να μιλήσω, αλλά δεν τα κατάφερα γιατί έχω μια ανησυχία για την έκθεσή του που έχει να κάνει με τα 45 λεπτά που είπε ότι μπορεί να είναι 3 φορές 15 λεπτά ανάπαυση. Εμένα μου δημιουργεί κάποια προβλήματα αυτά. Τέλο πάντων, διμερώ θα το δω με τον κύριο Βαντεκάμπ σε κάποια άλλη ευκαιρία. Τώρα, Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι το θέμα των χιλιόμετρων που χωρίζουν τους οδηγούς φορτηγών με τις οικογένειάς τους. Από το 2008 με την κρίση χιλιάδες νέοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και γυρνάνε μια-δύο φορές το χρόνο στα σπίτια τους. Λοιπόν, τον ίδιο ζήλο που δείχνουν οι χώρες που υποδέχτηκαν αυτούς με συμβόλαια ε, χαμηλών αμοιβών να δείξουν την ίδια ευαισθησία και για αυτούς όπως δείχνουν και για τους οδηγούς των ε, φορτηγών. Πονάει η καρδιά μου, πώς να σας πω. Να μιλάμε για κοινωνικές ευθύνες όταν πάρα πολλές οικογένειες, πολλοί από αυτούς τους νέους δουλεύουν αλλού και γυρνάνε στις οικογένειές τους αυτοί που μπορούν μια ή δυο φορές το χρόνο. Για αυτούς δεν μιλάμε, δεν μας ενδιαφέρουν, έτσι. Εκεί που υπάρχει ανταγωνισμός, με τη λιτότητα, βέβαια, οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, έτσι όπως έπεσαν οι μισθοί, είμαστε πιο ανταγωνιστικές. Και τώρα αρχίζουμε να νοιαζόμαστε για την ανταγωνιστικότητα. Τέλος πάντων, σχόλιο αυτό για να μην ακούω πια για αυτά τα κοινωνικά της ανοησίες μερικές φορές που ακούω και θα έρθω στα τόσο θετικά που λέει η κυρία Κιλόνεν. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για το ανοιχτό της πνεύμα, για τον νιάξιμό της για όλα αυτά τα θέματα και συμφωνώ μαζί της σε πάρα πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα, για τους ε, χώρους ανάπαυσης που λέμε ότι θα σταματάει ο οδηγός μάλλον όχι τους χώρους ανάπαυσης, συγγνώμη, ε, που θα γίνονται έλεγχοι στους δρόμους και θα σταματάει το φορτηγό και θα ελέγχεται στη μέση του δρόμου από τη στιγμή που θα γίνεται αυτό τεχνολογικά. Εγώ συμφωνώ μαζί της για το ότι αυτό πρέπει να γίνεται από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες πρέπει να συμμορφώνονται στο νόμο. Οπότε οι επιχειρήσεις πρέπει να ελέγχονται και όχι οδηγοί των φορτηγών. Αυτοί πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους. Άκουσα τι ζητούν τώρα οι συνάδελφοι που λένε ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια γιατί είναι σημαντικές αυτές οι δοκιμές για αυτούς. Έχω μιλήσει και με την Επιτροπή και την ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά της, για τη δημιουργικότητά της που με άκουσε και είπε κάτι που ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει τον έλεγχο με την τεχνολογία που έχουμε τώρα. Οι 60 ώρες κάθε 29 μέρες. Ίσως τότε θα μπορούσαν να γίνονται οι έλεγχοι αυτοί, οι μερικοί έλεγχοι. Πάντως βλέπω ότι η συγκεντρία δεν κατάφερε να καταλήξει μια συγκεκριμένη ιδέα. Προς το παρόν λοιπόν δέχομαι ό,τι λέει και θα δούμε. Μήπως υπάρξει δυνατότητα κάποια άλλη στιγμή να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Δεύτερον, Ευχαριστώ που δέχτηκε την πρωτοβουλία να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των ελέγχων τόσο στους αυτοκινητοδρόμους όσο και στις επιχειρήσεις. Για την ανταλλαγή πληροφοριών επίσης την ευχαριστώ πολύ και τους υπόλοιπους γιατί καταφέραμε να εντοπίσουμε αυτό το οποίο, για το οποίο μας βοήθησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να συμφωνήσουμε με τις αρχές. Πρέπει να ολοκληρώσετε τι είπατε? Λέω ότι πρέπει να ολοκληρώσετε. Α, να ολοκληρώσω, μάλιστα. Ε, δεν μου δώσατε χρόνο στην προηγούμενη συζήτηση, το παίρνω τώρα, γιατί εγώ είχα ζητήσει να πάρω το λόγο για να ρωτήσω κάτι τον κύριο Βαντερμπάκ, δεν μου το δώσατε, οπότε μιλάω τώρα. Λοιπόν, για την απόσπαση, συμφωνώ. Αν και με μερικά, δεν συμφωνώ απόλυτα για το καποτάς χωρίς απόσπαση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιάλα Σέντερ. Ο κύριος Λοτόφσκι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Κιλανέν. Ήταν πολύ δύσκολο το καθήκον του να εξευρεθούν συμβιβαστικές ε, τροπολογίες ε, σε αυτό το πακέτο για την κινητικότητα. Είναι σημαντικό που η συγγήτρια άκουσε τις απόψεις μας προσπαθώντας να τις συμφιλιώσει όλες παρά την ανελαίτη πολιτική πίεση ε, και μάλιστα τα καταφέρνει πολύ πέρα από την απλή πολιτική μεταφορών. Φτάνει στο χώρο της φιλοσοφίας και θέλω να την ευχαριστήσω γι' αυτό. Υποστηρίζουμε πλήρως την πιο πρόσφατη πρόταση με την οποία εξαιρούμε τις διεθνείς ε, μεταφορές και τις ε, διελεύσεις από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96 του. Είναι η μόνη λύση που θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε μια κρίση στον τομέα των μεταφορών. Επίσης δίνει τη δυνατότητα ανταγωνισμού σε όλες τις εταιρείες ε, Κάποιε λεπτομέρειε μπορεί να δημιουργούν ε, ανησυχίε, αλλά η γενική κατεύθυνση είναι πολλά υποσχόμενη. Ελπίζω ότι αύριο, καθώ θα συζητάμε όλα αυτά τα ζητήματα, θα καταφέρουμε να ε, αμβλύνουμε όλε τι διαφορέ και να βρούμε συμβιβαστικέ. Εξακολουθώ να μην συμφωνώ με την πολύ αυστηρή πρόσβαση στο οδικό σκέλος των συνδυασμένων μεταφορών. Σε αυτή την περίπτωση πράγματι η σχέση μεταξύ ε, των κανονισμών μεταφορών στις διάφορες χώρες ε, είναι σημαντική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το καμποτάζ και οι συνδυασμένες ε, οι πολυτροπικές μεταφορές αποφέρουν τεράστια ωφέλη για το περιβάλλον. Αν δυσχεράνουμε την συμμόρφωση με τους κανονισμούς αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις ε, και για τις απαιτήσει της κλιματικής πολιτικής. Στις σιδηροδρομικές και τις αεροπορικές μεταφορές ε, αναμφίβολα το άνοιγμα των εγχώριων αγορών έχει αποδώσει τεράστια ωφέλη. Ενώ αντιθέτω ε, δεν κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση στις οδικές μεταφορές. Αυτό είναι δύσκολο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ελπίζω λοιπόν ότι η θέση της Επιτροπής Απασχόλησης ε, που δεν μας φέρνει πιο κοντά σε συμβιβασμό δεν θα αποτελέσει παράδειγμα, δεν θα το ακολουθήσουμε. Ελπίζω εντός της Επιτροπής μας ε, να καταφέρουμε να βρούμε κάποια λύση φιλική προς τους οδηγούς ε, και φιλική προς τον κλάδο. Ευχαριστώ. Ε, τήρησα το χρονικό όριο, νομίζω. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σλατόφσκι. Κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κιλόνεν για τόσα είπε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που βάζει στο τραπέζι είναι τις αμφιβολίες και τις ερωτήσεις μας, τις καθημερινές, τουλάχιστον τις δικές μου, εμάς που έχουμε την ευθύνη τέτοιων εκθέσεων και γιατί έχουμε αμφιβολίες. Γιατί ήμουν πρόσφατα με συνδικαλιστές που μου έλεγαν ότι βλέποντας τις προτάσεις τροποποίησης, τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το χρόνο εργασίας και ανάπαυσης, ας μας αφήσουν καλύτερα όπως είμαστε τώρα, μου είπαν. Τι σημαίνει αυτό? Και εδώ συμφωνώ σε πολλά με την εισηγήτρια. Πρώτα απ' όλα, δεν καταφέρνουμε να εντοπίσουμε σωστά τα προβλήματα. Δεύτερον, η διαφοροποίηση που υπάρχει στην Ευρώπη καταστά την νομοθέτηση πολύ δύσκολο εγχείρημα σε μια δέσμη μέτρων όπως αυτό που έχουμε. Και το τρίτο είναι η κακιά μας συνήθεια στην πολιτική αλλά και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα η πολιτική μας αυτή η συνήθεια η κακιά να αναθεωρούμε όταν δεν έχουμε καταφέρει να εφαρμόσουμε σωστά τις προηγούμενες νομοθετικές μας αποφάσεις. Συμφωνώ το τον κύριο Μπαχ σε ένα πράγμα που είπε. Τι είπε. Είπε ότι θα βελτιωνόταν πολύ η κατάσταση αν εφαρμοζόταν σωστά η σημερινή νομοθεσία και αν κάνανε καλό έλεγχο οι χώρες μέλη. Και είναι αλήθεια αυτό, ισχύει. Αναθεωρούμε όλα αυτά τα μέτρα αντί να ζητήσουμε από τις χώρες μέλη να προβαίνουν σε έλεγχο και να εφαρμόζουν τα μέτρα. Και ποια είναι η λύση. Η εφαρμογή. Αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε. Ξέραμε ότι το καποντάζ ερμηνεύεται διαφορετικά στις διάφορες χώρες, ανάλογα με το που βρισκόμαστε. Γιατί δεν προσπαθήσαμε να λύσουμε αυτό. Τι εννοούμε όταν λέμε καμποτάζ. Για να καταλαβαίνουμε όλοι το ίδιο. Και αυτά σας τα λέω για να πω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε πως είναι περίπλοκη κατάσταση γιατί δεν ζητήσαμε το λόγο ευθύνε από αυτούς που τις έχουν. Δεύτερον, η συγγήτρια είναι αλήθεια ότι προσπαθεί να προβεί σε ένα άνοιγμα για να λύσει όλα αυτά τα ζητήματα που τίθεται και να είναι συνεπής και με τις άλλες οδηγίες για το καμποτάζ και το χρόνο ανάπαυσης. Μπορούμε να έχουμε ο καθένας την άποψή του, αλλά υπάρχει μια γενική συμφωνία για το ότι οι διεθνείς μεταφορές πρέπει να είναι εκτός αυτής της δέσμης μέτρων. Οπότε το ζήτημα είναι, μα περί τίνος πρόκειται τελικά, τι προσπαθούμε να ελέγξουμε την κινητικότητα των ανθρώπων, την κινητικότητα των επιχειρήσεων, την επιστροφή των οδηγών να γυρνάνε σπίτι τους, θα υποχρέσουμε κάποιον να επιστρέψει σπίτι του και να αυτός θέλει να πάει διακοπές. Τα λέω αυτά, γιατί είμαστε γεμάτοι αμφιβολίες όλοι, προσπαθώντας να αναθεωρήσουμε προς το καλύτερο την ομοθεσία Τέλος. Από τις νέες προτάσεις της εισηγήτριας, εμείς συμφωνούμε με πέντε. Χρειαζόμαστε περισσότερες εξηγήσει για τις δηλώσεις και για το θέμα των συνδυασμένων μεταφορών και αυτό σε συνδυασμό με το καποτάς. Οι τροπολογίες μας θέλουν απλοποίηση, νέες τεχνολογίες, δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας γιατί είναι ο μόνος κλάδος των μεταφορών που δεν έχει ευρωπαϊκή υπηρεσία και θα χρησιμεύε για την αναρμόνιση της νομοθεσίας, για τον έλεγχο και για την εφαρμογή ενός συστήματος όπως έχουμε για τους σιδηροδρόμους. Οι, οι έλεγχοι μάλλον στο καποτάς πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά και το θέμα των ευφυών ταχογράφων δεν μπορεί να περιμένει τόσο χρόνο. Αυτοί που θέλουν να επενδύσουν το κάνουν πολύ γρήγορα και έχει γίνει σε άλλους κλάδους, γιατί να μην γίνει και στις μεταφορές. Αυτά. Ευχαριστούμε. Η κυρία... Ευχαριστούμε κυρία Μπιλμπάου. Εγώ είμαι η επόμενη. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ ως κοιόδης θέλω να ευχαριστήσω για τις προσπάθειές σου προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία για ένα θέμα το οποίο δημιουργεί πόλωση και μην κρυβόμαστε, διαφοροποιεί τις διάφορες χώρες μεταξύ τους και τις διάφορες ιδεολογίες. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα βήμα με τροπολογίες που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της απόσπασης της διεθνείς μεταφορές. Όμω τελικά καταλήγουμε στο αντίθετο από αυτό που λέει η τελική δήλωση της Επιτροπής που προστέθηκε στον επίλογο μετά από τον τριμερή διάλογο βάσει της αρχικής οδηγίας του 96. Και σωστά γιατί τελικά η απόσπαση είναι μια εμπορική πράξη από κάποιον που προσφέρει υπηρεσίες σε έναν πελάτη μέσα στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή οι διεθνείς μεταφορές ε, εμπορευμάτων είναι ακριβώς αυτό. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι, τι σημαίνει αυτό. Αν βγάλουμε τις εμπορικές μεταφορές από αυτή τη ρύθμιση, αυτό θα ήταν μέγα σφάλμα και θα ήταν ένα πολύ ε, μεγάλο χτύπημα για την Ευρώπη. Το λέω δεν μπορούμε τους εργαζόμενους στις μεταφορές να τους συμπεριφερόμαστε σαν να είναι δεύτερης κατηγορίας. Δεν μπορεί να ξεχνάμε το ότι για ίδια δουλειά πρέπει να υπάρχει και ίδιος μισθός. Το αντίθετο σημαίνει ότι θα φτιάξουμε εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας με λιγότερη αναγνώριση, με λιγότερα δικαιώματα από τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι η ζούγκλα και άλλοι θα τρίβουν τα χέρια τους και θα λένε «Α, να, αυτό είναι η Ευρώπη». Ε, όχι, δεν είναι αυτό η Ευρώπη. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι σήμερα οι εργαζόμενοι στις μεταφορές πρέπει να προστατεύονται όπως όλοι οι μισθωτοί στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη δεν θα φτιαχτεί αλλά κάρτα. Βεβαίως και χρειάζεται πολύ θάρρος για να τίνουμε προς τα πάνω. Και για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε για ισότητα προς τα πάνω και όχι για μια Ευρώπη η οποία γίνεται όλο και πιο φιλελεύθερη. Ο καθένας βέβαια θα κάνει τις επιλογές του, αλλά οι συνέπειες δεν θα είναι ίδιες. Υπέβαλα τροπολογίες, γιατί κυρία Μπιλμπάο έχετε δίκιο. Το κοινωνικό dumping είναι αυτό που είναι. Μην ψάχνουμε για πράγματα που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει έλεγχο. Γι' αυτό και γίνεται κοινωνικό ντάμπινγκ. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ελέγχου. Δεν είναι δυνατόν για τι οδικέ μεταφορέ να μην υπάρχει. Δεύτερον, πρέπει, πιστεύω και το λέω καθαρά, η έλεγχοι να είναι ανοιχτοί και να μπορούν οι χώρες ε, μέλη να προβαίνουν σε τέτοιους. Πρέπει να υπάρχουν. Και τέλος, θα τελειώσω με τις τροπολογίες μου. Από την αρχή της μελέτης του, της δέσμης αυτής για την κινητικότητα, ε, πολλοί είπατε το ίδιο πολύ πήγατε επί τόπου, συζητήσατε με τους συνδικαλιστές, με τους δελικέριδες και τι μας λένε. Μας λένε ότι υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση, ότι υπάρχουν συνθήκες ζωής που θυμίζουν σύγχρονη δουλεία. Με αυτά τα λόγια. Η κινητικότητα πώς θα ανταλλάξει όλα αυτά για να μην υπάρχουν αύριο. Πρέπει όμως, γιατί αλλιώς εδώ θα τελειώσει το ευρωπαϊκό σχέδιο και δεν είναι αυτό που θέλουμε. Και πας περιπτώσει όσοι δεν έχουν φροντίσει για το αντίθετο να μην διαμαρτύρονται μετά. Ε, αρνούτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν αρνούμε τη βούληση της κυρίας εισηγήτριας ε, να επιτύχει συμβιβασμούς παρά τις πολιτικές ευαισθησίες όλες τις πολιτικές ευαισθησίες εκτός των εθνικών διότι όπως βλέπω αγαπάει τη χώρα της αλλά όχι όσο ε, ώστε να συμφωνεί μαζί μου. Τέλος πάντων, εκεί δεν είναι το πρόβλημα. Όσον αφορά όλα τα προβλήματα, το θέμα της απόσπασης των εργαζομένων σχετίζεται με την ε, υπηκότητα, όχι την πολιτική ε, ιδεολογία. Γι' αυτό λοιπόν οι φιλοευρωπαϊστές, ε, όχι Ευρωπαίοι, οι φιλοευρωπαϊστές ε, θέλουν να επεκτείνουν αυτή την αυτοκρατορία και να παραμείνουν πιστοί σε αυτή την πραγματικότητα. Αυτή η έκθεση και οι συμβιβαστικές δεν επιλύουν τα ουσιαστικά ζητήματα. Γιατί η εργασία ενός οδηγού αξίζει λιγότερο αφού πραγματοποιεί στην ίδια χώρα το ίδιο πράγμα που κάνει και ένα συναδελφός του από άλλη χώρα. Γιατί διότι η διαφορά μεταξύ των χρεώσεων επιτρέπει σε ορισμένους επενδυτές ε, να αποκομίσουν μεγαλύτερα ε, έσοδα, τόσο μεγάλα που όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση σοπά για να μην τους καταστρέψει και όσοι ξέρουν ότι θα αποκτήσουν ωφέλη κάνουν ότι δεν βλέπουν την αδικία. Η απόσπαση εργαζομένων έτσι όπως έχει σχεδιαστεί σήμερα επιτρέπει ένα πράγμα, την εκμετάλλευση ορισμένων εργαζομένων υπέρ κάποιων ανθρώπων. Και όλα τα υπόλοιπα παραμένουν σε δεύτερο πλάνο τελικά. Γιατί χάνουμε το ουσιώδε από μπροστά μα και τώρα με κάποιε τροπολογίε και κάποιε συμβιβαστικέ δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στο πρόβλημα. Πρέπει να καταργηθεί η απόσπαση των εργαζομένων, διότι αλλιώ θα καταργηθεί ολόκληρη ευρωπαϊκή ιδεολογία γιατί θα είναι το ίδιο με την εκμετάλλευση. Είναι δική μας ευθύνη και εμείς οι εθνικοί παρότι ξέρετε εγκαταλείπουμε την ιδέα της Ευρώπης γιατί, γιατί κατά την άποψή μας ε, είναι συμβίβαστη με την αξιοπρέπεια των φτωχότερων εργαζομένων οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενο εκμετάλλευσης ή βγαίνουν στην ενεργεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Αρνότου. Ζητώ συγγνώμη. Κυρία Λαμπάιεβα, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ναι, πράγματι είμαι ε, συντάκτρια της νομοδότητας της Επιτροπής Απασχόλησης. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για μένα προσωπικά ήταν μεγάλη απογοήτευση αλλά δεν θα πάψω να αγωνίζομαι για να πετύχω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και παρά αυτό που έγινε στην Επιτροπή μου, χαίρομαι πολύ που οι συνάδελφοι στην Επιτροπή Τραν γνωρίζουν πολύ καλύτερα τον τομέα αυτών και εκφράζουν απόψεις που αντικατοπτρίζουν την, πραγματικότητα. Ε, είχα διάφορες συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές ε, της Επιτροπής Τραν και ε, είχαμε πάντα ευρεία συνένεση σε όλες τις πολιτικές ομάδες και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κρυλώνεν που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και προσπαθεί να πετύχει ε, συμβιβαστικές προτάσεις ε, και ελπίζω πράγματι να καταλήξει σε συμβιβαστική λύση σε αντίθεση με αυτό που κάναμε στην Επιτροπή Απασχόλησης. Λοιπόν, η διαμετακόμιση ποτέ δεν θεωρήθηκε απόσπαση, δεν υπάρχει ε, απόσπαση στην χώρα διαμετακόμιση ε, διότι δεν φορτώνονται ούτε εκφορτώνονται προϊόντα εκεί. Θα πρέπει όμως να έχουμε σαφή αναφορά στον αποκλεισμό της ε, διαμετακόμισης στην πρόταση. Ενδομεταφορές. Πρότεινα και εγώ το ίδιο θέμα στην Επιτροπή Απασχόλησης, διότι υπάρχει ανταγωνισμός με τους εγχώριους μεταφορείς ε, διεθνείς μεταφορές. Ε, θα πρέπει να εξαιρούνται από τους κανόνες για την ε, απόσπαση. Αυτή ήταν η γνώμη μου ήδη από την αρχή και συνεχίζει να είναι η άποψή μου ακόμα και μετά το διαφορετικό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία. Και αυτό φαίνεται και στο σχέδιο γνωμοδότησή μου για την Επιτροπή Απασχόλησης. Και γιατί το λέω αυτό και γιατί νομίζω ότι θα είναι εδώ δύσκολος οποιοδήποτε συμβιβασμός, διότι ε, οι κανόνες απόσπασης ε, έχουν να κάνουν με, ε, λιγότερο κινητούς εργαζομένους, όπως είναι για παράδειγμα στον τομέα των οικοδομών. Είδαμε τρελά πρόστιμα, τρελές κυρώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Είχαμε απόφαση του δικαστηρίου της προηγούμενης εβδομάδας, όπου 8.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε σε αποσπασμένο εργαζόμενο επειδή δεν είχε στην, ε, στα γερμανικά τα ε, έγγραφά του στην Αυστρία οι κανόνες αυτοί περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν μιλάμε για τους κανόνες περί αμοιβής που βασίζονται στις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό θα είναι αδύνατο να εφαρμοστεί σε κάποιον που εκτελεί πολλές και πολύπλοκες επιχειρήσεις μεταξύ διαφόρων χωρών σε καθημερινή βάση. Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να μετράμε τις μέρες. Εγώ δυστυχώς πιστεύω ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει. Απλά ε, ξεχνάμε το πραγματικό πρόβλημα που είναι η εφαρμογή της οδηγίας περί απόσπασης. Έτσι κρυβόμαστε πίσω από τον αριθμό ημερών. Αυτό θα είναι εις βάρος κάποιων οικονομικών φορέων και επιπλέον η πρόταση υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασισμένη στην παλιά οδηγία. Τώρα όμως έχουμε νέους κανόνες και κανένας δεν έχει αξιολογήσει τις συνέπειες στον τομέα των μεταφορών. Νομοθετούμε στα τυφλά εδώ. Όσο δεν γνωρίζουμε το πραγματικό αντίκτυπο δεν θα πρέπει να διαμορφώνουμε κανόνες. Και τελευταία μου παρατήρηση, ε, θα πρέπει να θυμούνται αυτοί που διαπραγματεύτηκαν την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων υπήρχε σαφή σε συμφωνία να αναθεωρηθεί η μητρική οδηγία μόνο εάν διατυπωθούν συγκεκριμένοι κανόνες για τον τομέα μεταφορών. Θα πρέπει τώρα λοιπόν να σεβαστούν αυτή ε, την συμφωνία και όχι να αναθεωρήσουν την ε, τους κανόνες ε, της οδηγίας περί απόσπασης. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Απλά να πω ότι όπως φαίνεται αυτό το θέμα σε συνδυασμό με το καμποτάζ ε, εκεί βλέπουμε το χάσμα μεταξύ κρατών με μεγάλη ε, κοινωνική νομοθεσία και τα υπόλοιπα και σε σχέση όλα αυτά με την ανταγωνιστικότητα δημιουργούνται δύο μπλόκα συμβίβαστα μεταξύ τους Άκουσα προσεκτικά όλους τους ομιλητές και ανάλογα με την επικότητά τους ξέρω τι θα πούν. Χαίρομαι για την κινητοποίηση βέβαια της Ανατολής, είναι σημαντική και σας συγχαίρω. Ε, πολλοί μίλησαν, ε. Λοιπόν, η παρατήρησή μου είναι ότι συνδυάζονται τα δύο αυτά. Αν δεν υπήρχαν διεθνείς μεταφορές δεν θα χρειαζόταν να ρυθμίζουμε καμποτάζ, τελικά όλα θα ήταν ανοιχτά, θα καταστρέφαμε τα πάντα. Ε, αλλά να είστε βέβαιος, δεν θα συμβεί αυτό, διότι όπως ξέρετε στο Συμβούλιο τα πράγματα δεν θα γίνουν έτσι. Οπότε μπορούμε να προσπαθήσουμε αυτά που έχει γίνει σε άλλα θέματα της δέσμης ε, για την κινητικότητα, να βρούμε κάποια λογική λύση ή να βρούμε μια παράλογη. Ε, τελικά, κυρία εισηγήτρια ε, βγαίνοντας από τις ε, εθνικές από τις εθνείς μεταφορές και από το καμποτάζ ε, αυτό είναι ένα συμβασμός ξέρετε ότι είναι απαράδεκτο εντάξει μπορούμε να το ρισκάρουμε ψηφίζοντας ξέρουμε όλοι τι θα ψηφίσουν αλλά δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσει το θέμα και καλό θα ήταν να συνδυάσουμε όλα αυτά με το καμποτάζ ε, τέλος για τον κύριο Ντέλη διότι είναι ενδιαφέρουσα η σχέση που περιγράψατε για την επιστροφή των φορτηγών δεν είναι αθώο, είναι πολύ έξυπνο. Δεν ε, επιστρέφουμε τα φορτηγά. Τα φορτηγά παραμένουν εκεί, κάνουν το καμποτάζ και εμείς κάνουμε απλά εναλλαγή οδηγών. Με πουλμανάκια μάλιστα που έχουμε υποβάλει σε ειδικά μέτρα και αλλάζουμε τον κόσμο χωρίς να μετακινούμε τα φορτηγά, ούτε τα ρημουλκούμενα. Εγώ, ξέρετε, το έχω δει αυτό. Στη δική μου πόλη είχαμε τεράστια τα πάρκινγκ για φορτηγά όπου γινόταν η αναλλαγή προσωπικού το Σαββατοκύριακο. Για το Σαββατοκύριακο δεν μπορούσαν να κυκλοφορούν ώστε να συνεχίσουν να κάνουν καμποτάζ. Γι' αυτό το λόγο και τα φορτηγά πρέπει να γυρνούν πίσω. Αλλιώ εκεί έχουμε ένα σύστημα τελείω ε, ελεύθερο. Τι θέλω να πω με αυτό. Μην χάνουμε από τα μάτια μα ε, το σύνολο των μέτρων, το ε, δέσμη για την κινητικότητα, υπάρχει μια σχέση μεταξύ αποσπάσμενων εργαζομένων και καμποτάζ. Προφανώς πιστεύω ότι οι πιο ακραίες ε, μεταξύ εισαγωγικών προτάσεις ε, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουν τελικά σε κάποιο ρυθμιστικό μέτρο. Ε, οπότε πρέπει να τα σταματήσουμε από πριν. Οπότε αντί γι' αυτό ας προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάτι ισορροπημένο αντί να κάνουμε ατέρμονες συζητήσεις χωρίς κατάληξη. Ευχαριστούμε κύριε Ρικέ. Θα είμαι πολύ εύστηρη μαζί σας. Έχουμε ακόμα δύο εκθέσεις να εξετάσουμε. Έχουμε χάσει αρκετό χρόνο ήδη, οπότε προσπαθήστε να τηρείτε τα δύο λεπτά που σας δίνω. Ευχαριστώ κυρία Ταρπαντέλ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν ε, σε αυτή την εκθέση και σε όλες τις εκθέσεις που σχετίζονται με τη δέσμη για την κινητικότητα. Είμαστε ειλικρινείς εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών. Να σας ρωτήσω, εγώ ανέκαθεν συμφωνούσα ίση αμοιβή για ίση εργασία, αλλά τι κάνουμε με έναν οδηγό που αμείβεται από μια γαλλική ή μια γερμανική εταιρεία τον κατώτατο μισθό στη Γαλλία ή ακόμα χειρότερα τον κατώτατο μισθό στην Ρουμανία ε, όπου οι Γάλλοι είχαν μια εταιρεία γραμματοκιβωτίου ενώ ταυτόχρονα ο Γάλλος οδηγός που εργάζεται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα λαμβάνει πολύ μεγαλύτερη αμοιβή για την ίδια δουλειά. Τώρα όσον αφορά την οδηγία για την απόσπαση των οδηγών από τις πληροφορίες που έχω εγώ μετά από τη συνάντηση της 24 η Απριλίου φαίνεται η πλειοψηφία να είναι κατά του να συμπεριληφθούν οι μεταφορές σε αυτή την οδηγία. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η καλύτερη και πιο δίκαιη επιλογή. Γνωρίζετε ήδη τη θέση μου. Το να συμπεριλάβουμε τις διεθνείς μεταφορές ε, στην απόσπαση είναι θεμελιώδε λάθο, Θα οδηγήσει σε στρεβλώσει στην ε, αγορά μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας μην ξεχνάμε ότι το να συμπεριληφθούν οι διεθνείς μεταφορές αντίκειται και στην αρχή της ε, ίσης πρόσβασης στην ενιαία αγορά. Μιλάμε για πιο ανεπτυγμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ανατολικές και δυτικές. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Εδώ είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δίκαιο να ε, είναι μεγαλύτερος ο φόρτος για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό θα οδηγήσει στη που πολλών ε, μεταφορικών εταιριών. Με συνέπεια την απώλεια πολλών θέσεων εργασία, γιατί ε, πολλοί μεταφοροί στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη έχουν να υπολογίσουν όλε τι αμοιβέ όλων των οδηγών του ε, σε όλε τι χώρε από τι οποίε διέρχονται. Αντιλαμβάνεστε πόσο εξωφρενικό είναι αυτό. και κατά πόσο η κοινωνική η οικονομία, η κοινωνική οικονομία της αγοράς θα λειτουργήσει έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. να φτιάξουμε έναν Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τις Οδικές Μεταφορές είναι πολύ σημαντικό, καθώς και η υλοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Για δύο λεπτά, ε, επόμενος ομιλητής. Madame Κυρία Λουκάζοσκα, για δύο λεπτά. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τη Μύρια. Έκλεισε το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Ναι, σας ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Μύρια που προσπαθεί να βρει μια λογική συμβαστική πρόταση. Υπερασπιζόμενη τις επιχειρήσεις, τις θέσεις απασχόλησης και προσπαθώντας να βρει ε, συμβαστικά μέτρα εφαρμόσιμα στην πράξη. Ο κύριος Ερικέ είπε ότι δεν θα πρέπει να επιμείνουμε στις θέσεις μας. Δεν καταλαβαίνω. Έχω λάβει επιστολή από την γαλλική αντιπροσωπεία που λέει ότι επιμένει στην αρχική της θέση ε, και δεν θα δεχτεί τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι πνεύμα συμβιβασμού. Συμφωνώ με τους ομιλητές που λένε ότι ο τομέα αυτό δεν θα πρέπει να καλύπτεται από την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Αν έχουμε μια νοσοκόμα ή έναν ε, εργάτη οικοδομών ε, που πάει στην ε, Γερμανία ή τη Γαλλία, αυτή είναι τελείως διαφορετική περίπτωση από έναν οδηγό που περνάει μέσα από πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε δύο μέρες. Τι έγγραφα θα του δώσουμε για κάθε μισάωρο που περνάει από κάποια χώρα. Δηλαδή το μισάωρο που περνάει μέσα από το Βέλγιο θα αμείβεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λογικοί. Όχι μόνο για να μην γίνουμε ρεζίλοι ω ευρωβουλευτές, αλλά για να έχουμε και κανόνε εφαρμόσιμου στην πράξη. Θα πρέπει λοιπόν να απλοποιήσουμε την κατάσταση, να εξαλείψουμε τα ε, εμπόδια, να έχουμε ηλεκτρονικά έγγραφα και να καταπολεμήσουμε τις επιχειρήσεις βιτρίνα. Θα ήθελα όλοι μας να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε το, τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα, όχι μόνο υπό το φως της προστασίας των οδηγών, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ακούσαμε ότι η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Μακρόν θέλουν να προστατεύσουμε τον τομέα των μεταφορών αυτό με κάποιον τρόπο που να μπορέσει να αναπτυχθεί και να προστατεύονται οι θέσεις απασχόλησης ε, ε, θα πρέπει και ο καταναλωτής να πληρώνει το, το ανάλογο τίμημα. Ε, ευχαριστώ κυρία Ουρσκογκ. Θα μιλήσω σουηδικά. Αντικαθιστώ τον Γιάννη Νίλσον που έκανε εξαιρετική δουλειά ως μέλος της Επιτροπής μας. Ε, έχουμε ακριβώς την ίδια θέση με αυτή που παρουσίασε ο Γιένς Νίλσον ε, τα χρόνια που πέρασε στην Επιτροπή αυτή. Ε, πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε την σύγχρονη δουλεία στα πιο πλούσια μέρη του κόσμου, στην Ευρώπη δηλαδή. Δεν επιτρέπεται ο ανταγωνισμός προς τα κάτω, πρέπει να πετύχουμε ανταγωνισμό προς τα πάνω. συνάδελφος ε, Λουστρόφσκι είπε ότι ε, δεν ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το αποτέλεσμα της Επιτροπής Απασχόλησης. Οι δύο επιτροπές μας έχουν μοιρασμένη αρμοδιότητα στο θέμα αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να δεχόμαστε να αμείβονται οι άνθρωποι με τόσο χαμηλούς μισθούς και υπό τόσο κακές συνθήκες να λείπουν από το σπίτι τους επί μήνες. Πιστεύω ότι ο χρονικός περιορισμός των 48 ώρων ε, είναι αυτονόητο κατά τη γνώμη μου. Είμαστε από τις πλουσιότερες περιφέρειες όλου του κόσμου. Να μην μπορούμε να δεχτούμε χρονικό όριο 48 ωρών και να έχουμε ενιαίους κανόνες στις διεθνείς μεταφορές. Πόσο φτωχοί θα είμαστε αν δεν καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τάρενς δεν είναι εδώ. Ο κύριος Γκάρμπατσεφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα αστείο. Εάν πρέπει να επιστρέφουν κάθε τρεις, εβδο... κάθε τρεις εβδομάδες οι οδηγοί στο σπίτι τους, γιατί να μην ισχύει το ίδιο για τους ε, για τους ε, βοηθούς των ε, βουλευτών. Θα πρέπει και εκείνοι να μπορούν να επιστρέψουν σπίτι τους κάθε τρεις εβδομάδες να επισκέφτονται την οικογένεια τους και τους φίλους τους. Εν πάση περιπτώσει, είμαι μέλος της ομάδας σοσιαλιστών και δημοκρατών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιτρέπονται οι εντομεταφορέ και να έχουμε απόλυτα απελευθερωμένους κανόνες από ένα όριο και πάνω. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι γιατί είμαστε κατά της ε, ελευθέρωσης για τα φορτηγά ενώ είμαστε υπέρ όσον αφορά τα λεωφορεία και τα πούλμαν. Γιατί δηλαδή είναι τόσο κακό το καμποτάζ, οι ενδομεταφορές ε, στα φορτηγά, ενώ θεωρείται κάτι τόσο καλό όταν μιλάμε για τα λεωφορεία και τα πούλμαν. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ίσως επειδή οι επιχειρήσεις με ε, μεταφορές ε, αγαθών ε, εδρεύουν κυρίως στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, ενώ τα πούλμαν και τα λεωφορεία είναι κυρίως επιχειρήσεις της Δυτικής Ευρώπης. Ποιο είναι λοιπόν ο στόχος Μια τέτοια πρότασης. Προφανώς ο στόχος είναι οι επιχειρήσει από την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη να χρεοκοπήσουν και οι εργαζόμενοι τους τελικά να εργάζονται στη Δυτική Ευρώπη. Και αν δεν χρεοκοπήσουν να πρέπει να ξανακαταχωριστούν στη Δυτική Ευρώπη, κάτι που σημαίνει ότι οι πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης θα ε, πληρώνονται σε ταμεία της Δυτικής Ευρώπης και όχι της Ανατολικής Ευρώπης. Να σας συγχαρώ για αυτήν την αλληλεγγύη. Ε, δεν πρόκειται για αλληλεγγύη, ε, πρόκειται για απληστία. Ευχαριστώ κύριο Σκόχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι φυσικά πολύ που η η συγγήτρια θέλει οι έλεγχοι να γίνουν πιο απλοί και αποτελεσματικοί. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά το Lex Specialis, ας μην ε, ξεχάσουμε το σημαντικότερο. Θέλουμε πιο αποτελεσματική νομοθεσία, πιο εύκολα εφαρμόσιμη και πιο εύκολους έλεγχους. Θέλουμε επίσης θεμητό ανταγωνισμό στον τομέα αυτών, κάτι που δεν θα πετύχουμε με επιπλέον επιβάρυνση στις επιχειρήσεις μεταφορών. Αυτό θα το πετύχουμε μόνο αν βγάλουμε από την κυκλοφορία τα μαύρα πρόβατα όσον αφορά τις ενταμεταφορές. Ε, έχουμε άμεσο ανταγωνισμό με τις εγχώριες επιχειρήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται η οδηγία περί απόσπασης εργαζομένων. Όσον αφορά όμως την οδηγία τους διεθνείς, για τις διεθνείς μεταφορές θα παρακαλούσα την εισηγήτρια να ε, συνεχίσει να επιδιώκει πραγματικό συμβιβασμό. Δηλαδή ούτε εφαρμογή των κανόνων περί απόσπασης από την πρώτη ήδη ημέρα, ούτε μετά από δύο μέρες ή καθόλου. Θα πρέπει να βρούμε ένα μέσο ε, ώστε να πετύχουμε συμβιβασμό που να υποστηρίξει η πλειοψηφία. Ε, αυτή η μέση οδός, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν ε, τροποποίηση του ορίου που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή μετά από πέντε συναπτές ημέρες να ισχύουν οι διεθνείς κανόνες και οτιδήποτε ε, ξεπερνάει τις 9 ή 10 ώρες να ισχύει ως μία μέρα, να υπολογίζεται ως μία μέρα και οτιδήποτε λιγότερο να υπολογίζεται ως μισή μέρα. Αυτό λοιπόν ε, θα ήταν κάτι περισσότερο από ό,τι προτείνουν κάποιοι και κάτι λιγότερο από ό,τι προτείνουν κάποιοι άλλοι. Δηλαδή θα ε, πρόκειται για πραγματικό συμβεσμό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κόχο, κύριος Ερτούχ. Σας ευχαριστώ πολύ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ντίτερ Κοχ που πραγματικά καταβάλει προσπάθειες να διατυπώσει συμβιβαστική πρόταση ενώ όλοι οι άλλοι προλαλήσαντες ε, είπαν ότι ε, δεν δέχονται. Συνάδελφοι, όταν μιλάμε για απόσπαση εργαζομένων θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Βλέπουμε την κατάσταση που βλέπουμε στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους, διότι η νομοθεσία που ισχύει αυτή τη στιγμή επιτρέπει τόσα παραθυράκια που οι διάφορες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα εκμεταλλεύονται και γι' αυτό δεν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις στους χώρους στάθμευσης στους αυτοκινητόδρομους και ε, οι οδηγοί περνούν εβδομάδες μακριά από το σπίτι τους. Εάν λοιπόν θέλουμε να νομιμοποιήσουμε μια τέτοια κατάσταση Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ε, ε, θεσμοθετήσει το status quo χωρίς ε, να μπει στα χωράφια των κρατών μελών. Αλλά έχουμε υπερβολικά άνισες δυνατότητες εφαρμογής. Η Γαλλία και το Βέλγιο, για παράδειγμα, εφαρμόζουν διαφορετικά τους κανόνες από τη Γερμανία, η Γερμανία διαφορετικά από άλλες χώρες. Συνάδελφοι, ε, έχοντας υπόψη την πλειοψηφία της δικής μου πολιτικής ομάδας, ε, λέω ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε να αφαιρέσουμε συνολικά τις διεθνείς μεταφορές από την οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Ένα φορτηγό όταν αποχωρεί από ε, την χώρα καταχώρησής του και 365 ημέρες βρίσκεται εκτός της χώρας αυτής και πρέπει να επιστρέψει στη χώρα αυτή μόνο για τους ελέγχους. Ε, τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό συμφωνώ με τον Τίτερ Κόχ, θα πρέπει να βρούμε τη μέση εδώ Και αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα ε, και να τα ε, αντιμετωπίσουμε. Ε, δεν έχω άλλο χρόνο, θα κλείσω εδώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τελίσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ που είπατε, κυρία Πρόεδρε, ότι θα εφαρμόσετε τα δύο λεπτά. Θα έπρεπε να τηρείτε ο χρόνος ομιλίας, ξέρετε φοβάμαι ότι κάποιε από τι ακραίε θέσει για οποιοδήποτε από τα αρχαία αυτά, του φακέλου αυτού, θα έχει σοβαρέ συνέπειε, όχι μόνο στον τομέα των μεταφορών. Έχω και τη δική σα προσοχή, κυρία Πρόεδρε. βαριέστε από αυτά που λέω. Νόμιζα ότι είχαμε να κάνουμε με ένα ευαίσθητο ζήτημα. Έχουμε αμοιβαίο σεβασμό. Αυτά που λέτε... Μπορώ να κάνω δύο πράγματα συγχρόνως. Είμαι γυναίκα, ξέρετε. Δεν με ακούσατε θα μ' άρεσε να εφαρμόζετε τα δύο λεπτά από την αρχή και στον εαυτό σας ε, όταν δεν προεδρεύετε τη συνάντηση. Το δεύτερο, πρέπει σοβαρά να δούμε ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, συναγωνισμού μεταξύ επιτροπών ή μη ε, σεβασμού των κοινωνικών δικαιωμάτων. Το ζήτημα είναι ότι θα εφαρμόσουμε τις απόψεις της, ε, των, ε, των εργοδοτών αλλά οι μεταφορείς ε, ε εξυπηρετούν εμάς τις υπηρεσίες. Φαντάζεστε τι συνέπειες θα έχουμε. Δεύτερον, ας επιστρέψουμε στη ρίζα. Αν μου επιτρέπετε, ποιο ήταν το αρχικό πρόβλημα που εντοπίσαμε, από πού ξεκίνησε το πρόβλημα, το καμποτάζ. Οι ενδομεταφορές καταστρέφουν τις αγορές και εγώ το υποστηρίζω, διότι ναι, κάποιες από τις συμπεριφορές ορισμένων μεταφορέων δεν κάνω διάκριση μεταξύ μεγάλων, μικρών, ανατολικών, δυτικών. Ε, δεν χρειάζεται να ε, διαφωνούμε τόσο πολύ και να χωριζόμαστε από αυτού. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ε, οφείλεται στο καμποτάζ, όχι οι διεθνεί μεταφορέ, ούτε η διέλευση. Οπότε μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις διεθνείς μεταφορές και τη ε, διέλευση. Και θα πρέπει να δούμε και άλλους τομείς όπου υπάρχουν οι ίδιες συνέπειες και έτσι θα καταστρέψουμε την εσωτερική αγορά. Για μένα λοιπόν πρέπει να γίνει αυτό χωρίς διεθνείς μεταφορές, χωρίς διέλευση και να είμαστε αυστηροί και δίκαιοι από κάθε άποψη όσον αφορά το καμποτάζ της εταιρείας γραμματοκιβωτίου ε, τις πλασματικές δηλαδή εταιρείες, οτιδήποτε καταστρέφει τον ανταγωνισμό και την εσωτερική αγορά. Σκεφτείτε τις συνέπειες που θα έχουν ορισμένες διατάξεις, ορισμένες προτάσεις. Και εμεί θα είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Το ακριβέ, αποτέλεσμα θα το δούμε σύντομα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τέλισκα. Έχετε το λόγο κυρία Κυρία Βιέ. Ε, όπως είπε και ο συνάδελφος έχει σοβαρότατες συνέπειες για τις επιχειρήσεις και ξέρετε μιλάμε για γυναίκες και για άντρες και όπως είπε και η Μυρία, πρέπει να μην ξεχνάμε μια αρχή. Την, τον άγριο ανταγωνισμό μεταξύ Ευρωπαίων εργαζομένων ε, με αποτέλεσμα συνθήκες απαράδεκτης εργασίας που καταστρέφουν, όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, οποιαδήποτε αλληλεγγύη πολιτική στην Ευρώπη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το ζήτημα των αποσπασμένων εργαζομένων δεν μπορούμε να το αποκόψουμε από τη γενικότερη συζήτηση για τους αποσπασμένους εργαζομένους, δηλαδή τόσο τους οδηγούς όσο και τους υπόλοιπους ούτε να το βγάλουμε από το κοινωνικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από ισχυρότατη κινητοποίηση στον τομέα των μεταφορών που πλήττει την αξιοπρέπεια στο χώρο εργασία, το καθεστώ, την αμοιβή, τη υπηρεσία, και το βλέπουμε πολύ καλά στη Γαλλία, στην SNCF, στην Air France. Πιστεύω ότι η Γενική Οδηγία για την Απόσπαση Εργαζομένων κινείται προ αυτή την κατεύθυνση. Τόσο το καλύτερο. Αλλά Νομίζω ότι δεν μπορούμε να ζητάμε λιγότερα για τους αποσπασμένους εργαζομένους οδηγούς να λαμβάνουν την ίδια αμοιβή για την ίδια εργασία, να είναι ίσοι, ισότιμοι πολίτες. Τρία πράγματα επιβάλλονται. Η εφαρμογή του καθεστώτος απόσπαση εργαζομένων στις διεθνείς μεταφορές από την πρώτη μέρα. Αυτό υπόθηκε στη συζήτηση μέσω ρύθμισης αυστηρής του καμποτάζ και μέσω της ανάπτυξης ε, ελέγχων καθοδόν κυρίως. Και αυτό περιγράφεται. Ελπίζω οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν για αυτή την έκθεση να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αβιού. Στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κύριε Λεζό. Έχετε το λόγο κυρίως όσον αφορά το πτυχή της απόσπασης των εργαζομένων. Ευχαριστώ. είναι ένας από τους πιο δύσκολους φακέλους, ίσως όχι ο πιο δύσκολος, αλλά αρκετά ευαίσθητος για πολλές χώρες που έχουν εθνική νομοθεσία. Ένα στοιχείο που βγαίνει από τη συζήτηση είναι ότι χρειαζόμαστε σαφείς κανόνες για τις μεταφορές αυτές. Χρειαζόμαστε λέξεις specialis. Τώρα επί της ουσίας. Θέλω να υπενθυμίσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχει εδώ κάτι με το οποίο νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Είναι το καμποτάζ και το transit. Με την πρόταση της Επιτροπής θεωρούμε ότι ο ελάχιστος μισθός και απόσπαση πρέπει να ισχύουν από την πρώτη δραστηριότητα. Σε μερικές περιπτώσεις βέβαια το τρας είναι πάρα πολύ σύντομο, δεν ισχύουν οι κανόνες αυτοί. Τώρα επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της αρχής. Δεν θεωρούμε και δεν στηρίζουμε ένα σεβασμό που θα απέκλειε την εφαρμογή των κανόνων για το σας στις διεθνείς μεταφορές. Δεν πρέπει να υπάρξει τέτοιο συμβασμό και δεν θα γίνει μεταξύ των χωρών μελών. Χρειαζόμαστε βέβαια μια ισορροπημένη προσέγγιση και θεωρούμε ότι ελάχιστο ε, μισθός της απόσπαση προσφέρει ωφέλη στον ανταγωνισμό, αλλά είναι κάτι περιφερειακό αν το συγκρίνουμε με τις διοικητικές απώλειες. Και αυτό πρέπει να το πω για τον αριθμό ελάχιστων ημερών μετά από τις οποίες θα ισχύει αυτός ο μισθός. Είμαστε ανοιχτοί σήμερα να συζητήσουμε τις προτάσεις αυτές, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν στηρίζουμε να αποκλείεται η απόσπαση για τις διεθνείς μεταφορές. Τώρα για τις διοικητικές απαιτήσεις. Δεν συμφωνούμε ότι ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να είναι ανοιχτός για να επιλέξει ότι θέλει κάθε χώρα μέλος. Έχουν διαφορετικές απαιτήσεις όσον αφορά την απόσπαση και τις σχετικές δηλώσεις. Άλλος ζητάει να οριστεί ένας εκπρόσωπος. Αν δεχτούμε μια τόσο διαφορεπημένη προσέγγιση, ε, αυτό δεν είναι εσωτερική αγορά. Χρειαζόμαστε ένα περιορισμένο κατάλογο διοικητικών απαιτήσεων. Αυτό ήταν ε, το κυριότερο που ήθελα να σας πω σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λίζουα. Η κυρία Κίλωνεν για τα συμπεράσματα. Ως εισηγήτρια, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι πάντα ιδιαίτερη χαρά για μένα να ακούω πόσο εύκολος είναι αυτός ο φάκελος. Και έχω την αίσθηση ότι ό,τι και να κάνουμε, τελικά όλοι θα πεθάνουμε και ο πλανήτης θα καταστραφεί. Οπότε, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, δύσκολα θα είναι τα πράγματα. Θα συνεχίσω όμως το έργο μου με τους συνεργάτες μου, τους λαμπρούς, με τους σκιώδεις εισηγητές και θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε λύσεις. Λύσεις που να μας κάνουν να συνεχίσουμε να ζούμε δυστυχής μαζί για πάντα. Εξίσου δυσαρεστημένοι όλοι όμως, έτσι. Αυτά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κυρία Κίλονεν για αυτή τη θετική νότα που βάζετε. Ατομική και συλλογική, φαντάζομαι. Ωραία, υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 4 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με την έκθεση για το καμποτάζ και δίνω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ισμαήλ Ερτούκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, Όπως όλοι γνωρίζετε, λόγω του θλιβερού γεγονότος του θανάτου του συναδέρφου μας έπρεπε να αναλάβω το θέμα αυτό. Ε, έχω συνεχίσει τις εργασίες όμως στο πνεύμα των εργασιών του Γένς. Αύριο έχουμε την προς το παρόν τελευταία συνάντηση των σκιωδών εισηγητών και ήδη από την δεύτερη συνάντηση είμαι εισηγητής και προσπαθώ με τους συναδέρφους να συνεχίσω τις εργασίες πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, συναδέρφους ε, για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Μια σύντομη επισκόπηση για όσους ε, δεν ήταν παρόντες από την αρχή. Η Πράσινη φαίνεται να είναι η μόνη πολιτική ομάδα με ενιαία θέση στην ε, δεύτερη συνάντηση των σκιωδών ε, υπό την ε, δική μου προεδρία ασχοληθήκαμε με το θέμα της επιβολής του νόμου. Εξετάσαμε όλες τις τροπολογίες και καταφέραμε να πετύχουμε τη συνένεση όλων των πολιτικών ομάδων. Στην τρίτη συνάντηση ασχοληθήκαμε με τις κοινωνικές εταιρείες, εταιρείε γραμματοκιβωτίου ε, και συμφωνήσαμε πάνω στα μέτρα για να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο αυτό. Στην τέταρτη συνάντηση ασχοληθήκαμε με τα ελαφρά εμπαρικά οχήματα ε, στη, κατά την επόμενη συνάντηση τα κριτήρια για την πρόσβαση στην αγορά και νομίζω ότι πετύχαμε ε, καλά αποτελέσματα και με τη βοήθεια της γραμματείας μας. Η πέμπτη και τελευταία μέχρι στιγμής προς το παρόν συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο και θα ασχοληθούμε με τους κανόνες περί ενδομεταφορών. Και θα ασχοληθούμε και με το θέμα της ευθύνης. Θα ήθελα να σας ε, δώσω μια επισκόπηση των ε, συμβιβαστικών προτάσεων που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Όσον αφορά ε, την επιβολή του νόμου, στις 8 Απριλίου είχαμε τη σχετική συνάντηση. Οι πληροφορίες για τις αρχές ελέγχου θα πρέπει να είναι πλήρεις και διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο. Θα πρέπει να εναρμονιστούν τα εθνικά μητρώα και θα πρέπει τελικά όσον αφορά το προσωπικό, όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Έχουμε βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η συνεργασία με τις πιο σύντομες προθεσμίες για παράδειγμα όταν μια χώρα λαμβάνει αίτημα το οποίο αφορά άλλο κράτος μέλος. Ε, θα πρέπει η απάντηση να πραγματοποιείται όχι μέσα σε 10 μέρες όπως προέβλεπε η πρόταση της Επιτροπής, αλλά μέσα σε 5 μέρες. Επίσης, εάν ένα κράτος μέλος αρνείται ε, σε μόνιμη βάση να συνεργάζεται, ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία εις βάρος αυτού του κράτους μέλους και το διατυπώσαμε ως εξής «may take all necessary measures» μπορεί να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Προβλέπουμε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών ελέγχου καθώς και κοινά προγράμματα κατάρτισης κλπ. Όσον αφορά την ψηφιοποίηση, το ECMR, δηλαδή ε, η ηλεκτρονική φορτωτική και το θέμα του ταχογράφου συζητήθηκαν. και δίνουμε τη δυνατότητα εφαρμογής αυτών. Ο ΕΦΗ, ταχογράφος θα είναι υποχρεωτικό τουλάχιστον για τις διεθνείς μεταφορές και η ηλεκτρονική φορτωτική θα πρέπει να αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να ε, διατίθεται ήδη πριν ξεκινήσει η μεταφορά. Τα κράτη-μέλη επίσης ε, υποχρεώνονται να ελέγξουν την εφαρμογή. Όσον αφορά τις εικονικές εταιρείε. Ε, όσον αφορά τις εντομεταφορές και την απόσπαση, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικοί έλεγχοι και θα πρέπει να είναι δυνατή η ηλεκτρονική πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία. Θα πρέπει στην έδρα της επιχείρησης ε, να είναι ε, διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία και να επιτρέπεται και η ηλεκτρονική πρόσβαση στα δεδομένα αυτά στο κράτος μέλος όπου είναι καταχωρισμένα τα φορτηγά. Επιπλέον, ε, μια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό χώρων στάθμευσης ή μόνιμη πρόσβαση σε τέτοιες θέσεις στάθμευσης. Οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ, το ECR, κλπ. Ε, ήθελαν να είναι δυνατή η διάθεση των ε, ε, χώρων απασχολ... Ε, στάθμευσης και όταν είναι και με μίσθωση αυτών. Επίσης, θα ήθελα να περάσω στο... στην επόμενη ομάδα θεμάτων, τα ελαφρά φορτηγά και την πρόσβαση στην αγορά αυτών. Εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λύσουμε. Δύο λύσεις προτείνω εγώ ως εισηγητής. Είτε όλα τα φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων να συμπεριλαμβάνονται ή να καλύπτονται τα οχήματα από 2,5 έως 3,5 τόνους η πρόταση αυτή δεν είναι τόσο ευρεία όσο είναι η πρόταση της Κομισιόν να συμπεριλαμβάνονται όλα τα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων. Εγώ λοιπόν υποβάλλω αυτές τις δύο προτάσεις και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστική πρόταση που να μπορεί να υποστηρίξει η πλειοψηφία. Εάν η πλειοψηφία των πολιτικών ε, ομάδων στηρίξει την ε, πρόταση των οχημάτων 2,4 έως 3,5 τόνων, ε, τότε θα την προτιμήσω, ακόμα και αν γνωρίζω ότι το ΕΛΚ και το ECR θέλουν να συμπεριλαμβάνονται όλα τα οχήματα κάτω των 3,5 τόνων. Όσον αφορά τις διεθνείς μεταφορές, σημαντικό είναι το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ. Ε, για μένα αποτελεί σημαντικό συμβασμό το να περιορίσουμε τους κανόνες στις διεθνείς μεταφορές. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για τα ελαφρά οχήματα και το αργότερο 31 το δεκάτου του 2024 θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση για να έχουμε επισκόπηση της εικόνας στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους. Να γνωρίζουμε πόσα τέτοια οχήματα κυκλοφορούν. Αυτό αποτέλεσε αντικείμενο αντιρρήσεων διότι δεν γνωρίζουμε πόσα οχήματα κινούνται, ε, άρα το τι επιπτώσεις θα έχουν οι προτάσεις μας. Θέλουμε λοιπόν να συγκεντρώσουμε στοιχεία στο μέλλον για το θέμα αυτό. Όσον αφορά τα τέσσερα κριτήρια. Να υπάρχει εγκατάσταση σε κράτος μέλος, ε, να ε, έχει καλή φήμη η εταιρεία, η οικονομική κατάσταση της εταιρείας καθώς και η επαγγελματική ικανότητα συνεχίζουν να, να ισχύουν και για τα ελαφρά οχήματα, τα ελαφρά φορτηγά. Ε, έχουμε τους ε, λεγόμενους κοινούς, μικτούς στόλους, ε, δηλαδή μεγάλα και μικρά φορτηγά. Και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, την ερμανεύουμε ως εξής, ότι θα επιβαρυνθούν ανάλογα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, διότι θα πρέπει να διατηρούν ε, το ίδιο ποσό και για τα μικρά φορτηγά. Λέμε δηλαδή ότι για το πρώτο όχημα πρέπει να διατίθενται τόσα χρήματα, για το δεύτερο τόσα κλπ. Αλλά πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσει θα πρέπει να διαθέτουν μικρότερα ποσά για τα μικρά φορτηγά. Και φτάνουμε τώρα στο δύσκολο θέμα που είναι οι ενδομεταφορέ. Αυτό θα το συζητήσουμε αύριο. Το γραφείο μου έχει στείλει τις συμβαστικές προτάσεις και όπως σας είπα θα τις συζητήσουμε αύριο. Η πρότασή μου είναι να επιτρέπονται οι ενδομεταφορές σε ένα κράτος μέλος για 48 ώρες, δηλαδή τρεις μέρες. Ε, πρόκειται για δύο με τρεις μεταφορές ε, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο ανάπαυσης. Επίσης ε, προβλέπεται προθεσμία cooling off μέσα, χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο δεν επιτρέπονται για μεταφορές σε άλλο κράτος μέλος. Επίσης θα πρέπει να εξαρτάται από το εάν το φορτηγό έρχεται κατευθείαν από την χώρα καταχώρησής του ή ε, από άλλο τόπο. Επίσης, απαραίτητο είναι να επανέρχεται το όχημα στην χώρα καταχώρησης ε, προτού να επιτρέπονται οι μεταφορές. Για μένα και την πολιτική μου ομάδα και νομίζω και για πολλούς άλλους εδώ δεν ε, ε, αποτελεί θέμα συζήτησης όσον αφορά τις ενδομεταφορές ε, και την μη ύπαρξη εξαιρέσεων. Επίσης, το θέμα της ευθύνης δεν έχει ξεκαθαριστεί. Θα πρέπει να τιμωρούνται οι επιχειρήσεις ε, που ε, έχουν δώσει εντολή σε κάποιον που δεν τηρεί τους κανόνες. Πρόκειται για επίμαχο θέμα, το οποίο όμως θα συζητήσουμε. Αυτή λοιπόν είναι μια επισκόπηση των εργασιών αυτή τη στιγμή. Όταν διατυπώθηκε η νομοθεσία αυτή, και το ήλεγξα αυτό, οι ενδομεταφορές θεωρήθηκαν εθνικές μεταφορές και ε, προβλέφθηκε μόνο εξαίρεση ώστε να μην ε, ε, επιστρέφουν άδεια τα φορτηγά στην χώρα καταχώρησης. Ακούσαμε τώρα τη συζήτηση για τις αποσπάσεις και βλέπουμε κατάχρηση των κανόνων και γι' αυτό δεν μπορούμε να αφήσουμε τους κανόνες ως έχουν. Σας παρακαλώ λοιπόν να έχετε κατά νου ότι οι ενδομεταφορές είναι εθνικές μεταφορές, δεν έχουν να κάνουν με τις διεθνείς μεταφορές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ερτούγκ. Ανοίγουμε τη συζήτηση. Τρία λεπτά για τον καθένα. Κυρία Κασέσκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ λέει η κυρία Λουκασένσκα, ήθελα να ευχαριστήσω τον Ισμαήλ, καθώς και όλους τους συναδέλφους με τους οποίους συνεργαστήκαμε για το φάκελο αυτό. Όπως υπόθηκε ήδη, έχουμε επιτύχει συμβιβαστικές τροπολογίες για πολλά ζητήματα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος ότι καταλαβαίνουμε τους ορισμούς. Και πιστεύω ο καθένας μας αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει την επιχειρηματολογία των άλλων. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα μέχρι το υπεράτωση αυτού του φακέλου. Δεν θα επαναλάβω τα πράγματα επί των οποίων έχουμε συμφωνήσει όπως ε, για τους έξυπνους ταχογράφους και τα λοιπά ζητήματα τα οποία παρατίθενται εδώ κάναμε ό,τι μπορούσαμε ώστε να εξαλείψουμε οποιαδήποτε παρατυπία. Έχω μία αμφιβολία όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης. Είμαστε σε ένα σύγχρονο κόσμο. Δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις τα δικά τους οχήματα. Κάποιες τα μισθώνουν. Και οι χώροι στάθμευσης ε, δεν... Ε, ε, τους μισθώνουν. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουν δικούς τους. Οπότε και αναρωτιέμαι. Ε, αυτό. Και ήθελα να επανέλθω λίγο στις ενδομεταφορές στο καμποτάζ. Έχουμε λάβει συμβαστικές τροπολογίες. Ε, μάλιστα ακριβώς πριν μπούμε στην αίθουσα και δεν έχω προλάβει να τις κοιτάξω. Εκτενώς. Όσον αφορά την ευθύνη του επιμέρους κράτους μέλους, και το δίκαιο ανταγωνισμό και τον αθέμητο ανταγωνισμό, συγγνώμη. Αθέμητος ανταγωνισμός ο οποίος έχει αναφερθεί σε πολλές ε, ε περιπτώσεις και αναφέρεται ότι αν καλύψουμε το καμποτάζ με το κανονισμό απόσπαση εργαζομένων λέτε ότι αυτό θα οδηγήσει στην άρση οποιοδήποτε κοινωνικού dumping. Όπως φαίνεται από όσα ακούμε εδώ, οι περισσότεροι από εμάς Πιστεύουμε ότι το καποτάζ πρέπει να καλύπτεται από την νομοθεσία για την απόσπαση εργαζομένων από την πρώτη ημέρα. Στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο σημαίνει ότι από την ημέρα υπαριθμών 1 θα ακολουθούμε τους κανόνες του πλήρους ε, θεμητού ανταγωνισμού. Για ποιο λόγο να περιορίσουμε το καμποτάζ σε δύο μέρες λοιπόν αν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο δίκαιος ανταγωνισμός. Θέλουμε να έχουμε δίκαιες αμοιβέ ε, για τους οδηγούς και δεν θέλουμε να καταστρέψουμε και τον ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε το όριο των δύο ημερών. Αν το επιβάλλουμε αυτό το όριο των δύο ημερών, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να εξαιρέσουμε τους ε, πιο αποτελεσματικούς. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε από αυτού. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αρτούκ. Πιστεύω ότι αύριο θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ικανοποιητικές ε, συμβιβαστικές για όλους μας. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμά αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο είναι σημαντικό να καλυφθεί ε, το καμποτάζ από την πρώτη ημέρα από την νομοθεσία για την απόσπαση εργαζομένων και δεν πρέπει να έχουμε αυτό τον περιορισμό των δύο ημερών. Ίσως να υπάρχει κάποιο όριο, αλλά όχι δύο ημέρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λουκασένσκα. Κύριε Σλατόφσκι, έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για μια τόσο καλή δουλειά που έκανε και για την εξαιρετική οργάνωση των συνεδριάσεων των σκιωδών εισηγητών. Η ψηφιοποίηση, ο αγώνες για την καταπολέμηση των ψεύτικων επιχειρήσεων, όλα αυτά είναι θέματα που βάζουν πολλά ερωτηματικά. Αυτό που με τρομάζει εμένα πιο πολύ είναι ότι δημιουργούνται κάποιες συνθήκες πρόσβασης σε αυτή την αγορά και λειτουργίας του, που τελικά έχει επιπτώσεις και στην τιμή αυτών των υπηρεσιών και θα την πληρώσουν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα ελαφρά οχήματα για τις δικές τους μεταφορές, κάτω από τα, τους 3,5 τόνους δηλαδή. Είναι λοιπόν ε, πολύ σημαντικό το τι θα γίνει με τις οδικές μεταφορές, αλλά τι θα γίνει και με τις τιμές τους θα έπρεπε να βρούμε μια λύση η οποία να επιτρέπει να χρησιμοποιείται το καμποτάζ χωρίς νέους περιορισμούς και φραγμούς. Όσον αφορά άλλα συστήματα μεταφορών, δεν βλέπω γιατί να υπάρξουν δυσκολίες, γιατί η πρόσβαση στις αγορές αυτές είναι ανοιχτή σε όλους. Η χρήση των οδικών μεταφορών χρησιμοποιείται για πολλούς και διάφορους λόγους. Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η καταπολέμηση των καταχρήσεων αλλά δεν πρόκειται για ριζοσπαστικές αλλαγές που περιορίζουν ε, την αγορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επειδή αυτές δυσκολεύονται περισσότερο να τηρήσουν μια νομοθεσία ιδιαίτερα περιοριστική. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που τηρήσατε το χρόνο σας, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Τελίτσκα, εσείς τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ εκτιμάω το αποτελεσματικό έργο του εισηγητού και των συνεργατών του. Δεν θα μπορούσα να πω το ίδιο, παρόλο που καταλαβαίνω τις δυσκολίες, για τις συμβιβαστικές τροπολογίες που μας έφτασαν 24 ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Αυτά είναι δύσκολα ζητήματα. Πάντως η δυσκολία δικιά μου τώρα έχοντας ακούσει τον Ισμέλερ Τούκ και τους άλλους για την απόσπαση, είναι ότι δεν μπορεί κανείς να τα χωρίσει αυτά. Οι τοποθετήσεις για την απόσπαση και οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί για το καμποτάζ δημιουργούν μία εικόνα που δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία που να προσφέρει λογικές συνθήκες για την αγορά αλλά και να προστατεύει τα κοινωνικά δικαιώματα. Άκουσα τον κύριο Ερτούγκο και τον κύριο Βαντερκάπ που είπε πριν πως είναι σε διάθεση ε, συμβιβασμού αλλά κάποια στιγμή είπε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν επιδέχεται συμβασμό ε, τι στάση είναι αυτή. Τώρα, για το καμποτάζ, όπως είπα και πριν, είναι πρόβλημα. Η λύση είναι ακριβώς η καλή και λογική διαχείριση των διεθνών μεταφορών. Θα ήθελα να ξέρω τι θα περιορίσει το συστημικό καμποτάζ στην πρόταση αυτή. Δεν το εντόπισε, ίσως σε δεύτερη ανάγνωση να μπορέσω να το εντοπίσω. Έπειτα, σε τι βαθμό θα περιοριστούν τα προβλήματα αν το καμποτάζ περιοριστεί στη μία χώρα μόνο. Οι αγορές δεν είναι ίδιες αν έχουμε διεθνείς μεταφορές από μια περιφέρεια στην άλλη άκρη της Ευρώπης, γιατί δεν έχουμε διεθνή μεταφορά. Είμαστε σοβαροί με τους στόχους μας και τους περιβαλλοντικούς. Αν ναι, πρέπει να προσαρμοστούμε στην πραγματικότητα. Για μένα το θέμα είναι να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα και μετά να δούμε και την κοινωνική προστασία. Τέλο πάντων, θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί και ελπίζω να καταφέρουμε κάτι περισσότερο. Παραμένουν κάποια ζητήματα ανοιχτά, αλλά ελπίζω να καταφέρουμε να τα κλείσουμε και αυτά αύριο. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τελίσκα. Είναι η σειρά μου. Για το καμποτάζ, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Ισμαήλ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Ισμαήλ. Θέλω να υπογραμμίσω πρώτα απ' όλα ότι ο Ισμαήλ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ως εισηγητής. Κληρονομήσατε υπό δύσκολες συνθήκες το φάκελο αυτό. Το γνωρίζουμε όλοι. Αμέσως οικειοποιηθήκατε του θέματος εσείς, οι σκιώδεις και η γραμματεία σας βοήθησαν ώστε να περάσει στην Ολομέλεια πριν το καλοκαίρι όλο το πακέτο για την κινητικότητα. Αντιλαμβάνομαι, όπως βλέπω, Κάποιοι προσπαθούν να ξεφορτωθούμε οριστικά το καμποτάζ. Ωστόσο, δεν εκφράζεται κάποια τέτοια ανάγκη από το δικαστήριο. Σε μια πρόσφατη απόφαση για τη Δανία και την πολιτική της για το καμποτάζ, είπε το δικαστήριο ότι πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα η νομοθεσία. Διευκρινιστεί δεν σημαίνει να καταργηθεί ούτε να απογυμνωθεί από την έννοια της. Καθόμαστε και αναρχιόμαστε λοιπόν για τον περιορισμό του καμποτάζ ε, στι συνεδριάσει ε, εξέβρεση συμβιβασμών. Αύριο θα γίνει η τελευταία συνεδρίαση. Να υπενθυμίσω τι έγινε πριν από τρει εβδομάδε στην Επιτροπή Απασχόληση. Περιορίζοντα σε 48 ώρε ε, και μετά σε κάποιον αριθμό ημερών το καμποτάζ, η Επιτροπή έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα. Η απελευθέρωση του καμποτάζ δεν μπορεί να αποτελέσει λύση ενώ το φαινόμενο των οδηγών νομάδων αυξάνεται στους δρόμους μας με τρομακτικές κοινωνικές και οικονομικές ε, συνέπειες και με συνέπεια πολλά ατυχήματα. Ελπίζω ότι η Επιτροπή Μεταφορών θα έχει το πολιτικό θάρρος να υιοθετήσει παρόμοια θέση. Είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί η κοινωνική νομοθεσία σε θέματα οδικών μεταφορών και για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα Όλοι γνωρίζουμε σε αυτή την Επιτροπή, δεν είναι μυστικό, τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα είναι όλο και περισσότερα αντικαθιστούν τα βαρέα οχήματα σε διεθνεί μεταφορε εμπορευμάτων. Οπότε σα υπενθυμίσω, αγαπητοί συναδελφοί, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν θα αφήσουμε κανένα νομικό κενό. Θα εφαρμόσουμε τα τέσσερα κριτήρια σε όλα τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές. Το έχω ήδη πει, αλλά το επαναλαμβάνω. Έχει έρθει η ώρα να στείλουμε ένα χειρομήνυμα για το ζήτημα του κοινωνικού dumping. Δεν υπάρχει άλλη μέθοδος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχουμε έναν Ευρωπαίο χωροφύλακα, ο οποίος θα είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που θα διενεργεί πραγματικούς ελέγχους. Είναι απαραίτητο, διότι όσο ωραίους νόμου και να κάνουμε δεν εφαρμόζονται. Δεν μπορούμε τέτοια εποχή να λέμε θα εμπιστευτούμε τα κρατη Έχουμε δει τι γίνεται. Δεν θα επαναλάβω τώρα τι υποθέσει που ξέρουμε. Δεν έκαναν τίποτα. Οπότε χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό. Ευχαριστούμε Ισμαήλ. Ελπίζω να ληφθούν υπόψη τα όσα είπατε. Κυρία Κιλόνιν, έχετε το λόγο. Dear Chair, Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Ισμαήλ και την ομάδα του. Ε, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Νίλσον που βρίσκεται κάπου εκεί πάνω, κάπου εκεί ψηλά, έκανε κάποιες καλές αρχικές εργασίες που μας βοήθησαν και αυτό είναι το πιο σημαντικό πιστεύω. Μας άφησε ένα κληροδότημα σημαντικό. Καταφέραμε, πιστεύω, να συνεργαστούμε εξαιρετικά σε αυτά τα τρία πολύ δύσκολα ε, θέματα, την απόσπαση, το καμποτάζ ε, και τα οχήματα χωρίς οδηγούς και θέλω να ευχαριστήσω και το προσωπικό της Επιτροπής Τραν διότι συνεργαστήκατε μαζί μας πολύ αποτελεσματικά και πολύ συχνά ξεχνάμε να σας ευχαριστούμε. Έχουμε λοιπόν τώρα τις συμβαστικές τροπολογίες. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό στο τέλος ε, να βρούμε μια ε, καλή λύση με διάφορες ε, πληροφορίες που θα μπορέσουμε πραγματικά να εφαρμόσουμε, να αναγκάσουμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν μεταξύ τους και να μοιράζονται απαραίτητες πληροφορίες, για παράδειγμα για τους οδικούς ελέγχους και για τους ελέγχους των επιχειρήσεων. Εγώ με λύπη μου αντιλήφθηκα κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ότι μιλάμε για ψηφιοποίηση, έτος ψηφιοποίηση στην Ευρώπη, το γιορτάζουμε, κάνουμε διάφορα σεμινάρια για το πόσο ψηφιοποιημένοι είμαστε και τα συστήματά μας. Ενώ ουσιαστικά δεν συμβαίνει αυτό. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διάφορες λύσεις και πλατφόρμες ε, διαμοιρασμού πληροφοριών που είναι η βασική ανάγκη όπως και η εφαρμογή του υπάρχουσας νομοθεσίας. Ελπίζω λοιπόν να καταφέρουμε αύριο να βρούμε κάποιες λύσεις με ευθύνη δεν είναι εύκολο αλλά είναι πολύ σημαντικό Προτείνω επίσης και μια πλατφόρμα εμπιστοσύνης, όχι μαύρη λίστα. Πιστεύω είναι προτιμότερο. Να αναδεικνύουμε όσους κάνουν καλή δουλειά, να τους επενούμε και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούμε κίνητρα και για τους άλλους ώστε οι καλοί να έχουν κίνητρα να ακολουθούν τους κανονισμούς, να τους στηρούν και να κάνουν αυτό που πρέπει. Και έτσι θα αλλάξουμε την κατάσταση, τη ε, μορφή του ανταγωνισμού, αναδεικνύοντας ε, αυτό το θέμα ε, της καλής φήμης σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των οδικών μεταφορών. Το σημαντικότερο πιστεύω για εμάς είναι οι εταιρείε βιτρίνες, οι εταιρείε letterbox. Χαίρομαι που είμαστε πολύ κοντά στη λύση. διότι στον τομέα των οδικών μεταφορών αυτό είναι σημαντική συνιστόσα του δίκαιου ανταγωνισμού και δεν το έχουμε συζητήσει τόσο. Χαίρομαι λοιπόν που τώρα πλέον έχουμε τουλάχιστον την νομοθεσία στο μπροστά μας. Ευχαριστώ κύριε Κιλόνεν, κύριε Κόχ παρακαλώ. Για δύο λεπτά. Σε ευχαριστώ Ισμαήλ για την πολύ καλή δουλειά που έχεις κάνει όσον αφορά την πρόσβαση στην ε, απασχόληση και στην αγορά, ε, θα πρέπει να έχουμε συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού. Και αυτό θα το έχουμε εφόσον περιορίσουμε τις ενδομεταφορές, εφόσον δεν έχουμε ακόμα ενιαία αγορά με ενιαία φορολογία και συνθήκες πλαισίου. Επίσης, όσον αφορά το 48ωρο και την ε, και το χρονικό διάστημα cooling off και αυτά είναι απαραίτητα για μένα. Δεύτερον, εάν θέλουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής ε, ώστε να καλύπτει και τα φορτηγά ε, από 2,5 τόνους, θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις ε, με τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων. Τρίτον, η εγκατάσταση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει περιθώριο κατάχρησης ε, υπό τη μορφή εταιριών ε, γραμματοκιβωτίου, εικονικών εταιριών και θα ήθελα επίσης συμβιβασμό όσον αφορά το άρθρο 4. Και το κράτος μέλος εγκατάστασης και τις θέσεις στάθμευσης ε, άσχετα από το αν αυτές είναι ιδιοκτησία ή αν είναι μισθωμένες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κόχ. Πάμε στον κύριο Λοζουά, η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Άκουσα πολύ προσεκτικά τις εξηγήσεις του κυρίου Ερτούγκ για την εφαρμογή για τις ε, εταιρείες βιτρίνες συνολικά. Θεωρώ ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση στις εργασίες για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, τα LCV. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε δύο επιλογές. Η, την πρόταση της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία όλα τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα θα υπόκειται στους κανόνες πρόσβασης στο επάγγελμα. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε είναι ότι σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής θα εφαρμοστούν μόνο δύο από τις τέσσερις ε, συνθήκες για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Αν είναι να εφαρμόσουμε και τις τέσσερις συνθήκες για την πρόσβαση στο επάγγελμα και την υποχρέωση ε, κοινοτικής ε, αδειοδότησης θεωρούμε ότι το καλύτερο θα ήταν να ακολουθήσουμε τη δεύτερη επιλογή τότε που αναφέρατε τον Έχουμε τον κανόνα πρόσβαση στο επάγγελμα μόνο για όσους διενεργούν διεθνείς μεταφορές και για ελαφρά επαγγελματικά οχήματα από ε, μια χωρητικότητα και πάνω, 2,4 τόνους και πάνω. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, δεν θα σας κάνει έκπληξη αυτό που θα πω. Έχουμε ήδη εκφράσει άποψη μετά από το σχέδιο εκθέσης του κ. Νίλσον. Είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί. Ε, στα όσα λέτε. Θυμάμαι τη φιλοσοφία της προτέσης της Κομισιόν. Καμία απελευθέρωση, αλλά και κανένας περιορισμός. Προτείναμε ένα νέο κανόνα για το καμποτάζ, περιορισμένος αριθμός ε, ε, ε, διαδρομών σε πέντε μέρες. Μπορεί να θεωρείτε ότι είναι πολύ, αλλά εμείς θεωρούμε ότι 48 ώρες δεν είναι αρκετές. Είναι ένας περιορισμός σε σχέση με τη σημερινή νομοθεσία. Και όπως είπαμε ήδη, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάποιον τέτοιο κανόνα που να περιορίζει το καμποτάζ στις 48 ώρες. Παρομοίως, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα κανόνα που θα περιορίζει το καμποτάζ σε διαδρομές όπου το φορτηγό επιστρέφει ή έρχεται από το χώρο ε, ε, έδρας. Ε, ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους κοινωνικούς κανόνες στην έκθεση του κύριου Βαντεκάμπ. Δεν θα πρέπει να θεωρείτε... Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ένας φορε, μια εταιρεία να πραγματοποιεί καμποτάζ ένα διεθνές ταξίδι και όχι μόνο ο, κατά την επιστροφή. Κάτι τελευταίο για την περίοδο cooling off ήταν κομμάτι της πρότασης της Επιτροπής, είναι κομμάτι και μια συζήτηση που κάνουμε στο Συμβούλιο, ώστε να καταπολεμήσουμε το συστηματικό καμποτάζ. Όλα εξαρτώνται από τη διάρκεια αυτής της περίοδου cooling off. Αν μιλάμε για δύο-τρεις μέρες, μπορεί να γίνει δεκτό, αλλά αν η περίοδος αυτή είναι δέκα ημέρες για παράδειγμα, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Είναι ένας άλλος περιορισμός που δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λεζοά. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα, επενθυμίζω, στις 4 Ιουνίου στις 4 το απόγευμα. 4 Ιουνίου, 4 το απόγευμα. Συνεχίζουμε με την επόμενη έκθεση. Αλλά κύριε Στούκ, θέλετε το λόγο, λέτε. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Σύντομα. Τέθηκαν κάποια θέματα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε ο Βάβελ Τελίσκα, ο οποίος πιστεύει ότι αυτός ο συστημικός περιορισμός μάλλον που αναφέρθηκε στον ε, περιορισμό αυτόν, δεν υπάρχει περιορισμός για τις αναμεταφορές, υπάρχει ρύθμιση. Δεν είναι ακριβώς περιορισμός. Θέλουμε στο κάτω-κάτω αυτές οι αθέμητες ενδομεταφορές, το, αθέμικο, το αθέμητο καμποτάζ να ρυθμίζεται με νέα βάση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και όσον αφορά την απόσπαση ήδη από την πρώτη μέρα, είμαι ανοιχτό όσον αφορά τι διαπραγματεύσει, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ευρεία πλειοψηφία αριστερά και δεξιά υπέρ Ε, του να ισχύει ήδη από την πρώτη μέρα εντομεταφορών ε, η ρύθμιση περί απόσπασης. Και τρίτον, παρακαλώ, όλοι να σκεφτούν, αν έχουμε περιορισμό 48 ώρων, τότε ο αριθμός επιχειρήσεων, ο αριθμός μεταφορών δεν περιορίζεται. Δηλαδή μπορεί να κάνει κανείς όσες μεταφορές θέλει ή προλαβαίνει μέσα στις 48 αυτές ώρες και κατόπιν χωρίς περιορισμό να συνεχίσει τις διεθνείς μεταφορές. Δηλαδή, από τον τόπο Α ξεκινήσει η διεθνής μεταφορά και ήδη εκ των προτέρων έχει υποβληθεί ε, η ηλεκτρονική φορτωτική, η CMR. Έχουμε δηλαδή διεθνή μεταφορά από το Α στο Β. Στο Β έχουμε εκφόρτωση από αυτή τη στιγμή ξεκινάει το 48ωρο απεριόριστων ενδομεταφορών και εάν η επιχείρηση θέλει να συνεχίσει μετά με διεθνείς μεταφορές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κανένας περιορισμός. Το σημερινό πρόβλημα είναι όμως ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ε, τον, του παράνομου καμποτάζ. Μπορεί να πούμε μέσα σε 7 μέρες επιτρέπονται μέχρι 3 επιχειρήσεις μεταφορών, τρεις μεταφορές, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό δεν είναι εφαρμόσιμο, δεν μπορεί να ελεγχθεί. Γι' αυτό λοιπόν δίνουμε χρονικό περιορισμό και μπορούν να γίνουν όσες μεταφορές θέλει κανείς μέσα στο διάστημα αυτό. Η Κομισιόν λέει πέντε μέρες, εγώ λέω δύο και κατόπιν επιτρέπεται οποιαδήποτε διεθνής μεταφορά χωρίς κανένα περιορισμό και έτσι έχουμε ενιαία ώρα. Λέμε λοιπόν κάνετε όσε διεθνεί μεταφορέ θέλετε και δεν μιλάμε εδώ για απόσπαση, μιλώ για διεθνεί μεταφορέ. Δεν υπάρχει κανένα περιορισμό. Εάν όμω θέλω να μπω στην εθνική αγορά να κάνω τα μεταφορέ, τότε θα πρέπει να επιτρέπεται αυτό. Με περιορισμό όμως 48 ε, ε, ώρων. Οι εντομεταφορές είναι εθνικές μεταφορές, εγχώριε μεταφορές και όπως είπε ο συνάδελφο Κοχ, εφόσον δεν υπάρχει η ενιαία αγορά, εφόσον δεν έχουμε τα ίδια πρότυπα, τις ίδιες συνθήκες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να το ρυθμίσουμε έτσι, χωρίς, ε, χωρίς υπερβολικό κόστος. Και τελευταία πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να νομιμοποιήσει την ε, κατάσταση της άγριας δύσης που βλέπουμε στους αυτοκινητοδρόμους. Αυτό δεν θέλω να το δω ε, και γι' αυτό ε, προτείνουμε τις συγκεκριμένε προτάσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ερτούκ και περνάμε στην τελευταία έκθεση τα μισθωμένα οχήματα η κυρία Μοντέρο Ντεαγκιάρ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παρόντες εδώ, γιατί με την βοήθειά τους καταλήξαμε στις συμβαστικές μας προτάσεις. Θέλω επίσης να κάνω μια μικρή δήλωση όσον αφορά την δικιά μου την εμπλοκή και πώς δέχτηκα διάφορες προτάσεις που υποβλήθηκαν. Από πλευράς του ΕΛΚ, αλλά και προσωπικά εγώ, κάποιες τροπολογίες τις θεώρησα περιτές, γιατί αναφέρονταν σε κάποιες οδηγίες και σε κάποιους κανονισμούς που όπως λέω ήταν κάτι εντελώς περιτό. Υπήρχαν ήδη όλα αυτά τα στοιχεία. Εμείς προσπαθούμε από τις τελικές μας προτάσεις να επωφεληθούμε όσο γίνεται περισσότερο από οτιδήποτε μας καλύπτει όλους. Για την πρόταση τώρα πιο συγκεκριμένα θέλω να σας πω το εξής. Η πρόταση αυτή αναφέρεται στη, σε ένα άνοιγμα της ε, αγοράς για οχήματα μισθωμένα χωρίς οδηγό. από τη μία την άλλη χώρα μέλος. Από τη στιγμή που έχει καταχωρηθεί το όχημα, προφανώς και καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις και τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και έκθεση αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όταν μιλάει για την χρήση των μισθωμένων αυτών ε, οχημάτων για οδικές εμπορευματικέ μεταφορές, μας δίνει και κάποιες ενδείξεις, κάποια στοιχεία. Μιλάμε για πιο σύγχρονα οχήματα, έτσι, πιο οικολογικά, που ρηπαίνουν λιγότερο. Και μιλάμε για μια αγορά που θα σέβεται περισσότερο το περιβάλλον. Στόχος που μας ενδιαφέρει όλους. Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι οι επιχειρήσεις αυτές να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα για τις εμπορικές οδικές μεταφορές κάτω από τις ίδιες συνθήκες και όρους όπως συμβαίνει και με τα οχήματα που είναι σε άλλη χώρα μέλος. Χωρίς δηλαδή να δημιουργηθεί η παραμικρή διάκριση. Και να σας υπενθυμίσω ότι οι χώρες μέλη μπορούν να περιορίσουν την μίσθωση τέτοιων οχημάτων για τις εμπορικές μεταφορές από άλλη χώρα μέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που υπάρχουν, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι τέσσερις μήνες συνεχώς και δεν μπορεί να είναι πάνω από το 25% του συνολικού τέτοιου στόλου που διαθέτουν. Μέχρι τέσσερα οχήματα επίσης μπορεί να μισθώνει η καθετερία. Για να γίνει πραγματικότητα πάντως ο... το μέτρο αυτό, τα μισθωμένα αυτά οχήματα πρέπει να αποτελούν μέρος των ηλεκτρονικών οχημάτων, όπως αναφέρεται στην Οδηγία 1071 του 2009. Και είναι οι χώρες μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους που πρέπει να καταχωρούν τις ε, πληροφορίες για το που βρίσκεται αυτό το μισθωμένο όχημα, που κυκλοφορεί κλπ. Όλα αυτά πρέπει να τα δίνουν οι αρμόδιες αρχές. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι η διοικητική συνεργασία να γίνεται μέσω ενός ε, συστήματος ηλεκτρονικών ε, μητρών εσωτερικού, όπως προβλέπεται και για τους άλλους φακέλους της δέσμης κινητικότητας. Το τελευταίο μου σχόλιο έχει να κάνει με αυτό που καθορίζει τελικά την έκθεση αυτή. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι ένα έγγραφο το οποίο να επιτρέπει να αποφεύγουμε περί τα βάρη. Τόσο το Κοινοβούλιο όσο και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να μην νομοθετούμε χωρίς να αναγνωρίζουμε την πραγματικότητα ε, που ζουν στην καθημερινότητά τους οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις μας. Μας κατηγορούν ότι είμαστε μακριά. Οπότε εδώ αναφερόμαστε συχνά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε πρέπει να βρεθούν ε, μέτρα αναλογικής εφαρμογής χωρίς να γίνονται διακρίσεις σε βάρος ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτό όσον αφορά τις συμβαστικές προτάσεις τις οποίες καταλήξαμε. Ο κύριος Ρικέ, ωραία. Η κυρία Άντερσον που είναι η πρώτη σκιώδη εισηγήτρια. Παρακαλώ κύριε Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ πολύ τις προσπάθειες ε, της εισηγήτριας, ωστόσο δυσκολεύομαι κάπως με το θέμα αυτό, διότι υπήρξαν κάποια διαδικαστικά προβλήματα, αλλά και προβλήματα ουσίας. Γενικά, η θέση του S&D δεν έχει ληφθεί υπόψη στις συμβαστικές προτάσεις. Καταρχάς, όσον αφορά τη διαδικασία, είχαμε προβλήματα κατά τις συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Η τελευταία μεταφέρθηκε χρονικά την τελευταία στιγμή, το οποίο σημαίνει ότι διάφοροι δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν. Νιώθω ότι βιαζόμαστε και μάλιστα βιαζόμαστε διότι κανένας ε, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται πάρα πολύ, ενώ πρόκειται για πολύ σημαντικό θέμα. Θέλουμε λοιπόν ε, να πετύχουμε κάποια πολύ σημαντικά θέματα εδώ. Θέλουμε να έχουμε μια σωστή και δίκαιη αγορά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή δυστυχώ είναι η αρνητική μου παρατήρηση. Τούτου λεχθέντος νομίζω ότι έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο. Όσον αφορά τους περιορισμούς, το βασικό θέμα εδώ είναι τα κράτη-μέλη θα πρέπει για θεμητούς λόγους ε, δημόσιας πολιτικής να εφαρμόζουν ε, περιορισμούς σχετικά με την χρήση ε, ενοικιαζόμενων οχημάτων. Πολλές πολιτικές ομάδες λένε ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέγιστα όρια χρήσης ε, μισθωμένων οχημάτων, ε, ενώ η συγγήτρια λέει ότι πρέπει να υπάρχουν ελάχιστα χρονικά όρια. Και δεν απέχει πολύ απόστασή της από αυτή του Συμβουλίου, ε, αλλά εμείς απέχουμε πολύ από τη θέση του Συμβουλίου. Έχουν γίνει διάφορες προτάσεις και δυστυχώς καμία δεν φαίνεται πολύ ισορροπημένη. Δεύτερον, πολύ σημαντικό θέμα για μας και μάλιστα μόλις συζητήσαμε τώρα το θέμα των πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η νομοθεσία αυτή και οι παραβιάσεις ε, θα πρέπει να ε, επηρεάζουν το θέμα της καλής φήμης όσον αφορά το καμποτάζ. Ε, υπάρχει σχετική τροπολογία την οποία θα πρέπει να στηρίξουμε ως τμήμα βασικού συμβιβασμού όσον αφορά την επιβολή των κανόνων. Παρά τις εκκλήσεις μας στο θέμα αυτό δεν εισακούστηκαν. Επίσης, το θέμα αυτό δεν είναι κατά κύριο λόγο περιβαλλοντικό. Θα γνωρίζετε όμως ότι σύμφωνα με τη συνθήκη επιβάλλεται σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εφαρμόζουμε τις περιβαλλοντικές απαιτήσει σε ό,τι κάνουμε. Εμεί θέλαμε ένα όριο όπου να μην επιτρέπεται η χρήση παλαιότερων οχημάτων στο πλαίσιο αυτή τη νομοθεσία υποβάλαμε πρόταση 5 ετών. Ε, καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πολύ αυστηρό όριο και τα περισσότερα νέα οχήματα είτε είναι ελαφρά είτε είναι βαρέα ήδη συμμορφώνονται με τουλάχιστον ε, τα πρότυπα Euro 5 Θα θέλαμε λοιπόν συμβαστική πρόταση που να λέει ότι θα πρέπει να ε, ε, υπάρχει συμμόρφωση με τουλάχιστον τα πρότυπα Euro 5 και Euro 6, ε, οπότε φτάνουμε σε οχήματα παλαιότερα του 2009. Όσον αφορά την χρηματοδοτική μίσθωση, το leasing, το 93% των επιχειρήσεων στον τομέα αυτών συμμετέχουν στην Lease Europe, η οποία έχει δεσμευτεί για τη χρησιμοποίηση περιβαλλοντικών, περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι ο στόλος των οχημάτων ε, περιβαλλοντικά θα είναι πιο καθαρός, αλλά αυτό δεν προκύπτει από την νομοθεσία. Αυτό λοιπόν ε, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο. Και τέλος, σε πολύ σημαντικό θέμα για μας είναι ότι δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει διάταξη ε, περί, των δικαιωμάτων των εργαζομένων ή κοινωνικών προτύπων. Θα πρέπει όμως ε, να συμπεριλαμβάνατε κάτι για την κατάρτιση των οδηγών όσον αφορά τις γενικές απαιτήσει στην ε, χρηματοδοτική μίσθωση σχετικά με το όχημα που μισθώνεται, τον τρόπο μίσθωσης κλπ. Προτείναμε διάφορους τρόπους να το πετύχουμε αυτό, συμπεριλαμβανομένης τροποποίησης της οδηγίας σε σύπηση Επίσης προτείναμε ρήτρα για την κατάρτιση. Τώρα προτείνουμε άλλη συμβιβαστική πρόταση διότι κάποιοι θεωρούν ε, τον όρο κατάρτιση υπερβολικό. Εμείς λέμε απλά ενημέρωση τώρα πια, μια πολύ ήπια πρόταση. Καμία από αυτές τις προτάσεις όμως δεν ε, έγιναν αποδεκτές παρά λοιπόν τις τεράστιες προσπάθειές μας ε, και τα διαδικαστικά ε, θέματα που ανέφερα, που δεν είναι λάθο ούτε της γραμματείας ούτε τη συγγήτρια, δεν μπορούμε δυστυχώ αυτή τη στιγμή να δεχτούμε καμία συμβαστική πρόταση. Πολύ ευχαριστώ θα συνεχίσουμε το διάλογο. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ισχυρή επιθυμία να ψηφιστεί το θέμα αυτό την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την διαδικασία στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Άντερσον, κύριε Ντεμασμάκερ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια από βάθος καρδίας για την προσπάθειά της που ήταν ανοιχτή, διαθέσιμη. ώστε να καταλήξουμε στις συμβαστικές τροπολογίες. Σε γενικές γραμμές είμαστε θετικοί απέναντι στις συμβαστικές τροπολογίες. Για την ομάδα μας είναι κυρίως πολύ σημαντικό να υπάρχει ισορροπία. Από τη μια μεριά η ελεύθερη αγορά, από την άλλη μεριά η φορολογική πολιτική, η οικονομική πολιτική και η ε, πολιτική ασφάλεια των χωρών μελών. Η πρόταση λοιπόν πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτή ακριβώς την ισορροπία και για μας το κάνει. Τώρα η ελευθέρωση της αγοράς μίσθωσης των χωρών μελών είναι κάτι που πρέπει να αναπτυχθεί, να υπάρχει καλή καταχώρηση και συνεργασία βέβαια μεταξύ των χωρών μελών για την ομάδα μας. Το ECR αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι προτάσεις μας ελήφθησαν υπόψη και συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο. Ε, ίσως χρειάζεται κάποια μικρή προσαρμογή, εξού και θα στηρίξουμε μια τέτοια τροποποίηση. Πάντως θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αδέρφους και την εισηγήτρια για την καλή συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστούμε κύριε Τεμισμάκερ. Ο κύριος Φαμιδαμπόρου. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα λέει ο κύριος Μίλτεμπερκ. Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια της εισηγήτριας να καταλήξει σε μια ισορροπημένη κατά τη γνώμη μου άποψη όσον αφορά τα μισθωμένα οχήματα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μην έχουμε περιτούς περιορισμούς που εμποδίζει τους επιχειρηματίες ε, οδηγούς να κυκλοφορήσουν και να δραστηριοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα επίπεδο ελευθέρωσης των μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό. Δεν πρέπει να περιορίζεται η χρήση ε, τέτοιων οχημάτων ανα των 6 τόνων. Η συγγήτρια έχει υποβάλει τροπολογίες που εξακολουθούν εξακολουθούν να έχουν αυτόν τον περιορισμό. Στις διαπραγματεύσεις όμως, και πολύ χαίρομαι που βοήθησε σε αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πίστηκε με επιχειρήματα να μην υπάρχει πια ο περιορισμός αυτός. Έπειτα, ε, τα οχήματα αυτά πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται για τέσσερις συνεχείς ε, μήνες. για να αντιμετωπιστεί και υψηλή ζήτηση. Οι περιορισμοί πρέπει να είναι αναλογικοί. Στους συμβασμούς λοιπόν υπάρχει δυνατότητα περιορισμού με 25% όριο τέτοιων οχημάτων στο συνολικό στόλο οχημάτων της επιχείρησης. Συνεπώς πιστεύω ότι έχουμε καταλήξει σε ένα καλό συμβασμό. Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικές ομάδες που έχουν διαφορετική άποψη. Και αυτό είναι πρόβλημα γιατί θα πρέπει να είναι ε, ένας φακελός που δεν θα πρέπει να είναι επίμαχος γιατί είναι τεχνικός. Ενώ οι διάφορες ομάδες θέλουν να το κάνουν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πράγμα το οποίο περιπλέκει τα πράγματα και τον καθιστά πολιτικά επίμαχο. Έτσι θα χρειαστούμε και άλλους μήνες για να ολοκληρωθεί το έργο μας για την ε, δέσμη αυτή μέτρων κινητικότητας. Συνεπώς, επιμένω να υπάρχει ευελιξία από όλες τις πολιτικές ομάδες για να καταλήξουμε σε ένα τελικό συμβασμό και να υπερψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία ώστε να περάσουμε στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ Ματιό. Κυρία Βιού. Και εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ ποιοτική η δουλειά αυτή που έχει γίνει και που απομένει να γίνει. Δεν έχω πολλά να πω, θα επικεντρωθώ σε ένα σημείο. Το υπογράμμισα στην αιτιολογική σκέψη ότι πρέπει να ανοιχτεί η δυνατότητα μίσθωσης αυτοκινήτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων στην Ένωση και αυτό μπορεί να αποτελέσει βοήθεια στις επιχειρήσεις ε, για να αντιμετωπίζουν ε, ε, τυχόν προβλήματα στι δραστηριότητέ του, Ωστόσο, ενθαρρύνονται οι περιπτώσει απάτη και φορολογική και κοινωνική. Χρειαζόμαστε λοιπόν εχέγγυα. Οι συμβιβαστικές τροπολογίε όμως δεν γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση όπως έχουν προταθεί μέχρι στιγμή, Είναι ανεπαρκή. Εγώ από πλευρά μου υποστηρίζω και γι' αυτό υπέβαλα τροπολογίε, περιορισμό χρονικό και ποσοτικό το χρόνο της ενοικίασης το πολύ σε ένα μήνα δύο φορές το χρόνο και περιορισμό στο 27% του στόλου. Δεδομένων των συζητήσεων που γίνονται, εγώ θα ήθελα να αφιερώσουμε χρόνο να συνεχίσουμε να συναντιόμαστε και να συζητάμε ώστε να ε, γίνουν εκτενείς συζητήσεις. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας για να κινητοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω να ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Λιζό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η... Υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή. Αντίθετα όπω είπε ένα σκιωδή, οι συζητήσει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο κινούνται σε μεγάλο βαθμό προ την ίδια κατεύθυνση. Θα έλεγα δηλαδή ότι ο φάκελο αυτό μάλλον θα έχει σύντομο τριμερή διάλογο. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, υποστηρίζουμε το έργο του εισηγητή, όπως είπα, να αναφέρω συγκεκριμένα το νέο άρθρο 2 της πρότασης. Είναι πολύ σαφές, απλό ως αρχή, όταν ένας φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα όχημα στη έδρα του, στη χώρα έδρας του, μπορεί να το χρησιμοποιήσει οπουδήποτε ανεξάρτητα από πού είναι ταξινομημένο. Μόνο ένα σημείο ουσιαστικά θα θέλαμε να αλλάξει στο σχέδιο έκθεσης. Αναφέρθηκε ήδη από τον Σκιώδη αφορά τις ε, δραστηριότητες για ιδίο λογαριασμό. Δεν βλέπουμε για ποιον αντικειμενικό λόγο να περιορίσουμε αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Ε, μόνο τρία κράτη-μέλη ουσιαστικά ακόμα παλιωμοδίτικα θα έλεγα επιβάλλουν τέτοιους περιορισμούς μέσω της νομοθεσίας πέραν αυτού. Όπως είπα, υποστηρίζουμε πλήρως το σχέδιο εκθέσης αυτό. Δυστυχώς θα διαφωνήσω με τις θέσεις ε, ενός κοιόδους. Δεν βλέπω να υπάρχει λόγος να απαιτήσουμε από τους οδηγούς επιπλέον εκπαίδευση για τη χρησιμοποίηση καλύτερου οχήματος. Αν έχει κάποιο την άδειά του, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για το δικό του αυτοκίνητο ή αν νοικιάσει ένα καλύτερο. Οπότε το ίδιο ισχύει και για τους επαγγελματίες οδηγούς. Δεν βλέπω λόγο να υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσει λοιπόν για τα οχήματα. Είναι απαραίτητο αν δείτε το η μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν και τα νεότερα οχήματα είναι εντάξει και προωθούμε και τα περιβαλλοντικά θέματα εδώ. Βλέπετε πώς συνδέεται αυτό το κείμενο με το καμποτάζ, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε καχύποπτοι προς τους φορείς με καλύτερα οχήματα. Γιατί να τους υποπτευόμαστε ότι μπορεί να ε, πραγματοποιούν παράνομε δραστηριότητες. Δεν υπάρχει λόγος. Θα εκφράσω λοιπόν την υποστήριξη της Κομισιόν προς αυτή την έκθεση. Με μία επιφύλαξη μόνο να μην συμπεριλάβουμε εξαίρεση ή αυστηρότερη ε, μεταχείριση όσων πραγματοποιούν δραστηριότητες για ιδιολογριασμό τους. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο για να κλείσουμε. Η κυρία Μοντέρο, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι πήραν το λόγο από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Και θέλω να εκφράσω και την θλίψη μου για την στάση σκιωδών εισηγητών που ξαφνικά θέλουν να επιταχυνθεί η διαδικασία. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε αρκετό χρόνο και λυπάμαι γι' αυτό. Εξαιτία των κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μα ανάγκασαν να αλλάξουμε τη συνεδρίασή μα. Πάντω, καταφέραμε στι 8 το βράδυ να συναντηθούμε. Ήμασταν ε, όλοι, με εξαίρεση κάποιον, και μπορέσαμε να συζητήσουμε μια τεχνική Νομίζω ότι δέχτηκα τις περισσότερες τροπολογίες των σοσιαλιστών. Για άλλη μια φορά θα υπογραμμίσω το περιβαλλοντικό ζήτημα. Δηλαδή, κάθε όχημα το οποίο καταχωρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάποιες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Αυτό το είπαμε από την αρχή και προσπαθούμε να ενισχύσουμε οδηγίες που ήδη υπάρχουν. Όμως δεν θέλουμε να προσθέσουμε περιτά πράγματα. Όσον αφορά τώρα την κατάρτιση των οδηγών. Εδώ μιλάμε για μία έκθεση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό. Αυτή που έχουν ήδη καταρτιστεί, που έχουν ήδη δηλαδή άδεια, μπορούν να είναι κατάλληλοι να συμπεριληφθούν και εδώ. Εξάλλου, το 79 μπορεί και να ψηφιστεί χωριστά. Επιμένω ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει χωριστή ψηφοφορία. Τέλος, για τις συμβιβαστικέ ε, τροπολογίες δεν γίνεται μνήα ε, σε οχήματα 6 τόνων. Και θέλω να επιμείνω και να κάνω έκκληση να είμαστε λογικοί. Αν καθυστερήσουμε ακόμα περισσότερο, ε, τίθεται σε κίνδυνο όλα τα στοιχεία τότε. Έχουμε ένα έγγραφο που μπόρεσε να βελτιωθεί για κάποια ζητήματα και ελπίζω, ελπίζω να μην μπλοκάρουμε τα πράγματα. Μέχρι τώρα είχαμε μια καλή συζήτηση στις διάφορες συνεδριάσεις μας. Και εγώ έκανα πολλές υποχωρήσεις για να καταλήξουμε σε συμβασμό. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς. Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 24 του μηνός στις 9 στην επόμενη συνεδρίασή μας. 24 Μαΐου λοιπόν στις 9 το πρωί είναι η επόμενη συνεδρίασή μας. Για να ψηφίσουμε μεταξύ άλλων και σε αυτό. Καλό σας βράδυ.